Shall we start? Ladies and gentlemen. Shall we start? Thank you very much. Thank you. Good morning. Good morning. Um, can, if, can we adopt the agenda? Καλημέρα σας. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και έχω και κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω. Να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Έχετε όλοι και ένα αντίγραφο του newsletter ε, και ε, διαδικτυακά αναρτημένο αλλά και στο βάθος της αίθουσας. Εχθές το βράδυ έγινε μια συνεδρίαση με τους Προέδρους των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους 28 Επιτρόπους. Συμμετείχα φυσικά στη συνεδρίαση εκ μέρους ε, της Επιτροπής μας Εσωτερικής Αγοράς, προκειμένου να εξετάσουμε το σχέδιο εργασίας ε, για το 2015 και να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων από αυτού. Ο κύριος Γιούνκερ ε, ξεκίνησε τη συνεδρίαση και μετά ο κύριος Τίμερμανς παρουσίασε λίγο το πρόγραμμα και ήταν πάρα πολύ ε, συγκεκριμένος και είπε ότι το πρόγραμμα του 2015 πρέπει να είναι ακριβώς αυτό, ε, αυτό το οποίο σκοπεύουν να κάνουν το 2015 και όχι ό,τι σκοπεύουν να κάνουν για το 2016, το 2017, το 2017, αλλά μόνο τα του 2015 και όλα όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπήρχε υπήρχε τίποτα καινούριο. Εγώ στη συνέχεια έκανα μία ε, δήλωση συγκεκριμένη ε, για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εξετάσουμε τα πράγματα με ένα νέο ανανεωμένο τρόπο που ε, θα βασίζεται και στην καλύτερη νομοθεσία. Παρενέβην σε δύο ενότητες, ένα στη συζήτηση για την ενία αγορά και μία φορά στη συζήτηση για μια ε, καλύτερη εσωτερική αγορά με μια ισχυρή βιομηχανική βάση. Η ψηφιακή ε, ενιαία αγορά συζητήθηκε επίσης. Ε, υπήρχε παρέμβαση και από την Επιτροπή Πολιτικής, Πολιτικών Ελευθεριών για την προστασία των δεδομένων επί του θέματος. και επίσης από την Επιτροπή Πολιτισμού, όπου έγινε αναφορά φυσικά στα πνευματικά δικαιώματα. Η πρόθεσή μου δηλώθηκε σαφώς, είπα ότι μας ενδιαφέρουν βέβαια η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσης εργασίας, αλλά ε, με θέματα προστασίας καταναλωτή και κατά νου και φυσικά ε, έπρεπε να δούμε και τα, ε, την εφαρμογή μετά την νομοθεσία, να γίνει μια αξιολόγηση και γι' αυτό μετά τη θέση σε ισχύ της νομοθεσίας και θέλουμε να ξέρουμε ότι όλη η νομοθεσία θα έχει εξεταστεί και από ψηφιακή σκοπιά, όχι μόνο η νέα νομοθεσία, αλλά και η προηγούμενη θα πρέπει να προσ προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή και μάλιστα υπάρχει και η μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο η οποία ε, τονίστηκε και είναι ένας τομέας ο οποίος έχει δυνητικά ωφέλη και για την οικονομία μας και για τους καταναλωτές βεβαίως. και ήταν θετικά τα σχόλια για τις δηλώσεις αυτές και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κατόπιν, για την εννέα αγορά Ο κύριος Κατάινεν ε, έκανε την εισαγωγή στο θέμα αυτό. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ε, περισσότερης εμβάθυνσης της ενέας αγοράς και κυρίως στην εφαρμογή. Ε, και αυτά ήταν αυτά τα οποία ήθελα να θίξω και εγώ από πλευράς της Επιτροπής μας. Και ανέφερε επίσης και τη σημασία τη σωστή εφαρμογή τη ήδη συμπεφωνωμένη νομοθεσία, ε, ε, ε, την οδηγία για την εσωτερική αγορά, τι αλλαγέ στι δημόσιε συμβάσει, τα επαγγελματικά προσόντα, όλα αυτά τα οποία θα οδηγήσουν φυσικά και σε καινοτομία και υπάρχει και οδηγία για την καινοτομία και τα δικαιώματα του καταναλωτή. Όσον αφορά τη νέα νομοθεσία, οι διατάξεις ε, για την οδηγία για τις ε, ε, δημόσιες συμβάσεις και τις συμπερίληψη και της ενιαίας αγοράς στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ήταν κάτι το οποίο μας απασχόλησε. Και όλα αυτά φυσικά έλαβαν αρκετά θετικά σχόλια. Ξέρω ότι θα υπάρξει και ε, ψήφισμα για το ευρύτερο πρόγραμμα εργασίας, κατά πάσα πιθανότητα τον Ιανουάριο, από τις ομάδες. Ε, και αυτό που θα ήθελα να ξέρω εγώ είναι κατά πόσον εμείς θα, εφαρμοστούμε, ε, θα ασχοληθούμε με την εφαρμογή Μπορεί πρέπει να εξετάσουμε και εμείς ως Επιτροπή πώς θα παρακολουθήσουμε και θα είμαστε ενήμεροι για τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση της νομοθεσίας ε, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι συνέπειες είναι αυτές οι οποίες επιθυμούμε και δεν θα έχουμε και φυσικά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα με τους συντονιστές για να δούμε αν θα θέλαμε να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο από το χρόνο της Επιτροπής για να εξετάζουμε τις διαδικασίες εφαρμογής ε, και ε, να βλέπουμε πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα τώρα, να εγκρίνουμε τα πρακτικά της ε, προηγούμενης συνεδρίασης. Αυτό είναι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και αν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ε, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά και κατόπιν να περάσουμε στο σημείο 4, ενημέρωση σχετικά με τις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Να δώσω το λόγο στο συνάδελφο για να μας πει, στη συνάδελφο για να μας πει για τον τριμερή διάλογο για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, ε, επειδή υπάρχει διερμηνία στα τσεχικά, θα μιλήσω τσεχικά σήμερα. Έχω ένα καλά νέο να σας ε, διαβιβάσω. Μετά από δύο ε, τριμερείς διαλόγους και πάρα πολλές τεχνικές συνεδριάσεις τις οποίες ε, σας ανέφερα το Νοέμβριο, με χαρά μπορώ να σας πω ότι τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, είχαμε τον τρίτο και τελευταίο τριμερίο πολιτικό διάλογο ε, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εγκρίθηκαν οι πράξεις κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές ε, πράξεις για το άρθρο 6, παράγραφος 4 για την προστασία του προσωπικού και έγινε συζήτηση για το πώς θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια συμβιβαστική πρόταση, η οποία ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που παρουσίασε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό και φυσικά και τα υποστηρίξαμε. Στη συνεδρίαση αυτή ε, συζητήθηκαν και κάποιες εκκρεμότητες και θεωρώ ότι καταφέραμε να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούσαμε. Καταφέραμε λοιπόν να τηρήσουμε την εντολή η οποία δόθηκε και εδώ στην Επιτροπή και στην ε, Ολομέλεια. Θέλουμε να έχουμε δωρεάν υπηρεσία ανεξάρτητα από το σύστημα που διαθέτουμε και αυτό το σύστημα, το λεγόμενο alert σύστημα, πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη και να βελτιώσει όλες ε, ε, την ασφάλεια συγγνώμη, στα οδικές μεταφορές. Ζητήθηκαν κάποιες περαιτέρω προθεσμίες από τα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω ότι αυτό που είχε σημασία για μας είναι να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η υπηρεσία. Η υπηρεσία η οποία προϋποθέτει να υπάρχει και διασύνδεση μεταξύ των ενδιαφερομένων, να είναι αποτελεσματική βεβαίως και να λειτουργεί ε, χωρίς προβλήματα. Ήταν ε, παρόντες φυσικά και οι συγητές από την Επιτροπή Μεταφορών και την Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών και θα ήθελα εδώ επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω την πρόοδο διότι επικεντρωθήκαμε σε πολύ συγκεκριμένα θάματα στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου και ε, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαπραγματευτική ομάδα και τους κοιόδης συγητές αλλά και τους βοηθούς, τους πολιτικούς συντονιστές, τη γραμματεία. και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιταλική Προεδρία για την εξαιρετική και παραγωγική συνεργασία. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα το υποστηρίξει η Επιτροπή μας αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ, Όλγα. Ευχαριστώ όλη την ομάδα διαπραγμάτευσης και τη γραμματεία για όλα όσα μπορέσατε να πετύχετε. Αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε στο συμφωνημένο κείμενο στις 10 σαν επιτροπή θα γίνει η ψηφοφορία και ελπίζω ότι από εκεί και πέρα θα υποβληθεί η θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο ελπίζω να ακολουθήσει την ε, ίδια διαδικασία με το κείμενο και τελικά θα επανέλθει το κείμενο στην ε, Ολομέλεια έτσι ώστε να ψηφιστεί. Τι να σας πω, πιστεύω ότι πριν την τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Κορεπέρ θα μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό κείμενο. The next Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι views um, uh, just one announcement. Το θέμα των εγκαταστάσεων με σειρματόσκηνα. Ε, υπάρχει εδώ ένα θέμα με τα κείμενα, τα μεταφρασμένα. Ε, εδώ βεβαίως πρόκειται για σχέδια εκθέσεων και εννοείται να ευχαριστώ τον Άντωνη είναι διαθέσιμα μόνο στα ισπανικά και στα αγγλικά προς το παρόν τα σχέδια εκθέσεων στις 11 Δεκεμβρίου και συζήτησα με την γραμματεία για το εάν η προθεσμία αυτή 11 Δεκεμβρίου για την υποβολή τροπολογιών θα πρέπει να παραταθεί ως οι σκιώδεις εισηγητέ με τους εισηγητές θα πρέπει να συζητήσουν και να πάρουν την απόφαση για το θέμα αυτό. Έχεις το λόγο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, μέχρι τώρα εργασία σου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συμφωνώ. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες ε, επιφυλάξεις και ανησυχίες για την έκθεση αυτή. Θα περιμένουμε να δούμε εξάλλου πότε θα είναι διαθέσιμες οι μεταφράσεις και περνάω στα ισπανικά. Η αγορά των εγκαταστάσεων με σειρματόσχηνα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εξειδικεύσης. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, έχουμε κάνει αυτή την έκθεση που είναι κατεξοχήν τεχνικού περιεχομένου για το οποίο υπάρχει πολιτική συνένεση. Η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το 60% της παγκόσμιας αγοράς αυτού του είδους των εγκαταστάσεων και μιλούμε για 4.000 θέσεις εργασίας που έχουν άμεση σχέση με τις εγκαταστάσεις μεταφοράς με σειρματόσχηρα. Η οδηγία του 2000 είναι το νομικό πλαίσιο, 2009 οδηγία 2009 που θέλει να αντικαταστήσει με κανονισμό η Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω την πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου ότι πρόκειται για παράδειγμα εναρμόνιση τη κοινοτική νομοθεσία. Με την πρόταση αυτή θέλουμε να εναρμονίσουμε τι συνθήκε που ε, επικρατούν ώστε να μπορέσουν στην αγορά να υπάρχει ασφάλεια στα θέματα εγκαταστάσεων με σειρματόσχηνα, υποδομές, υποσυστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας. Ένα από τα προβλήματα τα οποία εντοπίσαμε με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας 2000 ήταν το θέμα της διαφοράς στην μεταφορά σε εθνικές νομοθεσίες. Γι' αυτό πιστεύω το ότι όταν περάσουμε από την οδηγία σε κανονισμό θα έχουμε την πολιτική συνένεση να εργαστούμε σε όλα τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρχει εναρμόνιση και απλοποίηση των διατάξεων. Επίσης θα πρέπει να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ε, ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη χάρη στην εναρμόνιση δεν μπορούν ε, στην εθνική τους νομοθεσία να κάνουν κάτι λιγότερο ή περισσότερο από αυτό που προβλέπεται. Άρα θα συνεχίσουν να είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις με σηματόρφινα, καθώς και με θέματα που είναι χωροταξικά ή αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να μην έχουμε συμπληρωματικό κόστος από τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, θα έχουμε κάποιους κανόνες που θα ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επίση είναι κάτι το οποίο κατά τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία μας ε, προστατεύει από διαστευρώσεις στην εθνική αγορά και από αποκλήσει σε θέματα εφαρμογής. Πράγμα το οποίο δεν μας αρέσει. Στις διάφορες τροπολογίες που κατέθεσα κάνω τις διάφορες προσαρμογές όσον αφορά ε, την ε, μεταφορά των προϊόντων και συνεχίζω την εργασία την οποία έκανε η Επιτροπή μας και ε, κυρίως προσαρμόζομαι στην πρόταση 768-2008. Η πρόταση έκθεσης σέβεται την ε, διατύπωση την οποία είχαν ακολουθήσει οι συνάδελφοι που είχαν νομοθετήσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Και λαμβάνω υπόψη τα θέματα της εναρμόνισης έτσι όπως αναφέρονται στην Οδηγία 29 του 2014 για την εναρμόνιση. Προτείνω διάφορες τροπολογίες για να βελτιώσω την συνεκτικότητα του κειμένου στα πλαίσια του νέου νομοθετικού πλαισίου. Καταρχήν είχε προβλεφθεί διάφορες διατάξεις για ε, επαγρύπνηση στην αγορά σε θέματα ε, μεταφοράς με σειρματόσια να είναι παραμφερής με αυτά τα οποία γίνονται για την μεταφορά εμπορευμάτων, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό. Δεδομένου ότι δεν θα μπορέσει να εγκριθεί έγκαιρα αυτή η πρόταση, για διάφορα θέματα επαγρύπνησης στην αγορά έχουν προβλεφθεί νέες προτάσεις και προτείνω να προβλεφθεί η προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου 4 για θέματα ασφαλείας στην αγορά και για διασφάλιση των εγγυήσεων που μπορούμε να δώσουμε στην νέα αγορά. Εδώ δίδεται απάντηση στα θέματα της εφαρμογής της οδηγίας 2000 Παύλα 9 για την μεταφορά ατόμων. Καταρχάς η μελέτη επιπτώσεων εξάντε είχε αποφασίσει ότι θα πρέπει ένας από τους αντικειμενικούς μας στόχους να είναι η βελτίωση της σωστής νομικής βάσης και νομικής ασφάλειας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει οι διάφορες εταιρείες που κάνουν αυτού του είδους τις μεταφορές ε, που διαθέτει τις εγκαταστάσεις των συρματώσεων, τις υποδομές και τα υποσυστήματα, καθώς και τα καταστηματικά ασφάλεια, ασφάλειας για να λειτουργούν αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις με ασφάλεια, να σεβαστούν αυτές τις διατάξεις και καλύπτονται εδώ και τα άτομα τα οποία μεταφέρονται για εμπορικούς λόγους και η χρησιμοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων για λόγους ψυχαγωγίας. Αυτό δεν συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν για λόγους ψυχαγωγίας στα λούνα πάρκε τους παρεμφερείς χώρους ψυχαγωγίας. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη επίσης να εγγυώνται ένα υψηλού επίπεδου ε, σύνολο κανόνων ασφαλείας και για όλους όσους ε, αλλοδαπούς και πολίτες κάθε χώρας χρησιμοποιούν για λόγους ψυχαγωγίας αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις. Κατά την άποψή μου, τα υποσυστήματα επίσης θα πρέπει, καθώς και τα κατασκευαστικά συσχεία ασφαλείας, να τα ε, εξετάσουμε βάσει των ιδίων κανόνων και να προβλέψουμε την ίδια μεταχείριση για να μην υπάρχουν, όπως είπα και προηγουμένως, στρεβλώσεις στην αγορά. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας θα πρέπει, έτσι όπως προβλέπεται σχετική οδηγία, να λειτουργούν με ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, εδώ γίνεται και μία ε, νέα επανεκτίμηση, ώστε όλα να γίνονται βάσει των κανόνων που προβλέπονται στα νέα νομοθετικά πλαίσια. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο παρέλειψα. Παρακαλώ τους συναδέλφους να κάνουν παρατηρήσεις ώστε να συνεισφέρουμε στο να παρουσιαστεί μία πολύ καλή ε, έκθεση για το θέμα αυτό που είναι τόσο ώρα. Ευχαριστώ. Οι συγγητές, οι σκιώδεις, δεν ξέρω ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Λούσι Άντερσον από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την πάρα πολύ λεπτομερή και ε, σαφέστατη παρουσίαση αυτής της, ε, του σχεδίου έκθεσης. Όσον αφορά την ε, προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, θα ήθελα να προτείνω το εξής. Πρόκειται για μια ημερομηνία δύσκολη, γιατί είναι ακριβώς πριν τις διακοπές. Θα ήταν καλό λοιπόν εδώ να το επιμηκύνουμε λίγο αυτό το χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τώρα το θέμα του κανονισμού σε σχέση με την πρόταση για οδηγία, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε πολύ πιο συνεκτικοί και να λάβουμε υπόψη μας ότι εδώ υπάρχουν και θέματα επικουρικότητας για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να προτείνουμε ακριβώς αυτό που αρμόζει. Όπως προτείνει λοιπόν εδώ ο εισηγητής θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, να αποσαφινιστούν και να εναρμονιστούν σε ένα σημαντικό βαθμό όλες αυτές οι ρυθμίσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις για που αφορούν σειρματόσκηνα και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να κατανοήσουμε το φάσμα και το εύρος ενός ε, κανονισμού. Επίσης είναι πολύ σημαντικό εδώ ο ορισμός ε, κάποιων πολύ συγκεκριμένων ε, όρων να γίνει όπως παραδείγματο χάρη το θέρμα της συμμόρφωσης των φορέων και οργανισμών συμμόρφωσης, υποπτίας όπως ορίζει το άρθρο 15. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό κάποιες πληροφορίες να εγγράφονται στην συσκευασία, να υπάρχει δηλαδή σαφέστατη ε, επισήμανση και ετικετοθεσία. Θεωρώ επίσης ότι ουσιαστικά εδώ με αυτό το κανονισμό προσπαθούμε να επεξεργαστούμε το θέμα. Πρόκειται για θέματα ασφάλειας, πρόκειται για θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε πολύ πιο συνολικά. Και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας όσον αφορά την αναγραφή κάποιων πληροφοριών στη συσκευασία. Ξέρω ότι τουλάχιστον στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ενωμένο Βασίλειο, η αρμόδια επιτροπή έχει εξετάσει όλες αυτές τις ρυθμίσεις και για το τι ίσχυε πριν από το 2004 και αυτό που θεωρούμε πολύ σημαντικό είναι ήδη αυτά που υπάρχουν να εφαρμόζονται ορθά. Το θέμα λοιπόν των ιστορικών εγκαταστάσεων με σειρματόσχηνα όπως τις ονομάζουμε δηλαδή οι εγκαταστάσεις που εξαιρούνται είναι πάρα πολύ σημαντικό να οριστούν με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Παραδείγματος χάρη σε κάποιους σιδηροδρόμους, σε κάποιες παλιές εγκαταστάσεις, αυτό που ονομάζουμε ιστορικές εγκαταστάσεις με σειρματόσημα, δηλαδή θα πρέπει να οριστούν με πάρα πολύ ακρίβεια. Θεωρώ λοιπόν ότι λίγος παραπάνω χρόνος θα ήταν πολύτιμος και χρήσιμος. Ευχαριστώ πολύ, ECR. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Λόπες Ιστούρου, τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την Νίκη. Θεωρώ ότι ο χρόνος εδώ είναι απαραίτητος. Υπάρχει μόνο αγγλικά και ισπανικά η έκθεση αυτή και είναι μια πολύ συγκεκριμένη και τεχνική έκθεση. Θα χρειαζόμασταν λοιπόν ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και ένα κείμενο στη γλώσσα μας για να το εξετάσουμε γιατί χρειάζονται κάποιες τεχνικές γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το θέμα της νομικής βάσης για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει εδώ να μειώσουμε τις πιθανότητες περαιτέρω νομικών θεμάτων που θα προκύψουν αν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης ε, βλέπουμε ότι χρειάζονται πολύ συγκεκριμένοι ορισμοί, αποσαφήνιση κάποιων ορισμών όπως το θέμα των ιστορικών εγκαταστάσεων με σηματόσχηνα. Για την Άλδε, ο Τίτο Τράζ. Ευχαριστώ. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. 141 τροπολογίες. Τι παραπάνω να προσθέσω εγώ. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πολιτικών ομάδων για το θέμα αυτό. Το θέμα των ιστορικών εγκαταστάσεων και των εξαιρέσεων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, να το προσέξουμε. Στην Τσεχία έχουμε τέτοιες ιστορικές εγκαταστάσεις και σαφώς και θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, περί τίνος πρόκειται. Παρόλα αυτά και αυτές οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι ασφαλείς για τους χρήστες. Αυτές λοιπόν οι εξαιρέσεις θα πρέπει να μην οδηγήσουν σε επιπλέον καταχρήσεις, γιατί πολλές εγκαταστάσεις θα θελήσουν να ενσωματωθούν σε αυτή την κατηγορία των ε, ε, ιστορικών ε, εγκαταστάσεων γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξοικονομηθούν κάποιες δαπάνες επιπλέον ε, για τους ιδιοκτήτες. Το θέμα της εποπτείας, της επιτήρησης της αγοράς επίσης είναι πολύ σημαντικό, όπως μας περιγράψατε στα εισαγωγικά σας σχόλια. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια τεχνικά θέματα θα ήθελα εδώ να ρωτήσω την Επιτροπή όταν υιοθετηθεί ο κανονισμός για την εποπτεία της αγοράς, όταν συμφωνήσουμε για τους κανόνες αυτούς, τελικά αυτές οι ρυθμίσεις στον κανονισμό αυτό και την εποπτεία της αγοράς ε, υπερέχουν των διατάξεων αυτού του κανονισμού. Ερώτηση κάνω προς την Επιτροπή. Επίσης θεωρώ ότι δεν υπάρχει ανάγκη για οδηγία, υπάρχουν πολύ λίγοι αν θέλετε που παράγουν, πολύ λίγοι κατασκευαστές σε λίγα κράτη-μέλη, άρα μπορεί πολύ εύκολα να ευθυγραμμιστούν εδώ με τα πρότυπα τα οποία θα θεσπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Δεν θα κάνω εδώ συγκεκριμένε προτάσεις. Απλώς γενικότερε ερωτήσει θα ήθελα να θέσω όσοι συζήτηση για την ε, κανονισμό ασφάλειας γενικότερα των πρωτεόντων και σκιώδηση συγγήτρια για την ασφάλεια στην αγορά. Θα πω ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, ένα δυνητικό πρόβλημα, διότι μιλάμε για εγκαταστάσεις με σειρματός, να έχουμε και άλλου είδους ε, ε, φακέλους παρεμφερείς που αφορούν θέματα ασφαρούν και είναι μέρη του πακέτου ασφαλείας τα προϊόντα. Πώς θα μπορούμε να ασχοληθούμε και να λύσουμε το πρόβλημα αυτό της ασφαλείας. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε στο Συμβούλιο να ενεργήσει σε θέματα ασφαλείας, να προχωρήσει το όνορφάκι, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε και στην Επιτροπή μας. Πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε να ενεργήσουμε ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε του ίδιου επίπεδου προτάσεις, υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές και τους ε, διανομής αυτών των ανθρώπων καταναλωτή και τους κανονισμούς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι τέτοιοι ότι κυρίως σε θέματα εποπτείας της αγοράς θα έχουμε υποχρεώσει, οι οποίε θα είναι παρεμφερεί. για να μην έχουμε διαφορετικού κανόνε και κανονισμού. Αυτό είναι κακό για την ενιαία εσωτερική αγορά και δεν είναι καλό για κανένα. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε αυτό το οποίο θα ήθελα να υποδείξω είναι όντω να έχουμε με την νομική υπηρεσία μια συνάντηση για να συζητήσουμε το πώ μπορούμε να χειριστούμε το θέμα αυτό. Και ω Επιτροπή θα ήθελα επίση να πω ότι θα πρέπει να το θέσουμε και στο Συμβούλιο. Υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να ενεργήσουμε με κάποιο τρόπο ώστε να μην έχουμε πέντε ή έξι διαφορετικές νομοθετικές ε, ε, πράξεις, αν ε, θα πρέπει να έχουμε μια, ένα οριζόντιο πακέτο ασφαλείας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς πρέπει να ενεργήσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι κάνουμε θα είναι ορθό. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε, θα πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, η, επιτροπή, Γραμματεία της Επιτροπής έχει εξετάσει τους τρεις ε, ε, φακέλους που αφορούν τις ε, εγκαταστάσεις, τα σειρματόσχηνα, τις υποδομές, τα υποσυστήματα στα πλαίσια του νέου νομοθετικού πλαισίου για να δει πώς θα μπορέσουμε συνεκτικά για καθένα αυτά τα θέματα να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να σιγουρευτούμε το ότι η γραμματεία της Επιτροπής μας θα έρθει σε επαφή και με όλους αυτούς που αφορούν με το πακέτο ασφαλείας για να δούμε αν μπορούμε ε, όλοι μαζί από κοινού να καταλήξουμε σε μία συμφωνία για αυτό το είδους τα θέματα, ώστε να κάνουμε κάτι το συνεκτικό στην προσέγγιση μας. Όχι μόνο για τους κατασκευαστές επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τους εισαγωγείς και τους κατασκευαστές τρίτη χωρών, ώστε σε θέματα εποπτείας της αγοράς να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Θα ήθελα τη δική σας σύσταση να την φέρω στην γραμματεία για να δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέτε. όλα αυτά όμως νομίζω ότι ήδη έχουν κάνει πολύ προπαρασκευαστική δουλειά. Η Μαρίνα Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το γεγονός ότι παρουσιάστηκε σωστά αυτή η έκθεση. Πιστεύω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών όχι μόνο για αυτή την έκθεση που είναι πάρα πολύ πολύπλοκη αλλά γενικά δεν είναι μεγάλη αυτή η προθεσμία που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε όντως πολύ περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε και να σκεφτούμε τα θέματα αυτά, διότι νομοθετούμε για 28 χώρες και η ευθύνη είναι μεγάλη. Δεν ξέρω αν κατάλαβα κάτι λάθος, πρέπει να με ενημερώσετε. Συμφωνώ ότι όντως ότι στην ε, αντικατάσταση της οδηγίας 2009 με κανονισμό υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν είναι ε, πλήρως σαφή. Στο άρθρο 2 για τις, εγκατα... για τις εγκαταστάσεις με σηματών για τη μεταφορά προσώπων στα Λούνα Πάρκ και στα πανηγύρια κυρίως όσον αφορά τους τουρίστες, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να προωθήσουμε τον τουρισμό, όπως ξέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι πρόκειται για μια οικονομικά πολύ επικερδή δραστηριότητα. Στη Ρουμανία, στη χώρα μου, Φερρυπίν, Έχουμε τους κανονισμούς και δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδικό κανονισμός σε κάθε χώρα χωριστά, γιατί ίσω μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε στην έκθεσή σας λοιπόν ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία για τις τουριστικές αυτές εγκαταστάσεις όσον αφορά την μεταφορά προσώπων με τα σηματόσχηνα τι έχουμε και με τι θέλουμε να τα αντικαταστήσουμε όλα αυτά για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και η Κάθριν Στάιλερ τώρα, αλλά πριν μιλήσει η Κάθριν, δεν μου έδωσε κάποιο όνομα ασχεδόν από την ΚΟΕ, τους Πρασίνους, το EFTD. Αν υπάρχει κάποιος σκιώδης, ναι, από ό,τι φαίνεται Μπορώ να δώσω κάποιον, σε κάποιον το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ Βίκη. Από πλευρά των Πρασίνων εγώ έχω την τιμή να είμαι σκιώδης ε, εισηγητή για την έκθεση αυτή. Να πω ότι ε, αυτή τη στιγμή καταρχάς ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Δεν έχω ακόμα εξετάσει τις 143 τροπολογίες, ζητώ συγγνώμη, αλλά ε, εμπιστεύομαι τους συμβούλους της ομάδας και θα το κάνω και ε, να σας πω ότι ε, θεωρούμε ότι ε, πρέπει να τεθούν αυτά σε εφαρμογή και φυσικά ο εισηγητής μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη των πρασίνων για το έργο του και για τις προθεσμίες που έχει θέσει και για το γεγονός ότι ασχολούμαστε με αυτόν τον κανονισμό. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της παράλυσης που υπάρχει στο Συμβούλιο όσον αφορά τον εγκάρσιο και οριζόντιο χαρακτήρα του θέματος της ασφάλειας. Απλώς πήρα το λόγο λοιπόν για να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι γενικώ συμφωνούμε. Thank you, Madam uh, Chairwoman. Η κυρία Στάιλερ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όσους ασχολήθηκαν με αυτά τα θέματα και ξέρουμε ότι είναι πολύ αριθμό. Όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, θα μιλήσω και κάποια στιγμή για το αέριο. Και ε, ξέρετε ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στα θέματα εποπτείας της αγοράς είναι αυτές οι προτάσεις ε, ε, διότι εμείς θεωρούσαμε ότι είχαμε αντιμετωπίσει το θέμα της εποπτείας αγοράς και τελικώς βρισκόμαστε ενώπιον αυτής της καινούργιας πρόκλησης, διότι εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε υποστηρίξει κάποια συγκεκριμένα πράγματα από πλευράς Επιτροπής μας και τώρα έχουμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το ΕΛΕΦ, αλλά υπάρχει και δική μας η άποψη. Το να προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία ε, είναι ένα πρόβλημα. Ο εισηγητή, ο κύριος Αρντεμόζα, έχει δίκιο ε, για την εποπτεία τη αγορά και... Ε, ναι, μεν είναι ακαθόδε το ζήτημα, διότι έχουμε βρεθεί ενώπιον αυτή τη κατάσταση. Δεν το έχουμε επιλέξει εμεί, αλλά ε, μπορούμε να βρούμε το σωστό τρόπο να το λύσουμε το ζήτημα. Και ήδη το γεγονό ότι υπάρχει κάποιο που ασχολείται με το θέμα και ε, ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για το θέμα αυτό. Χαιρόμαστε που έχουμε και την ε, πρόεδρο που έχει την έκθεσή τη. Εγώ έχω την άλλη έκθεση και ο κύριο Λόπεθ Στουρίθ ε, White έχει την τρίτη έκθεση και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνέπεια και στα τρία αυτά ζητήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Μάρκος Πρέτσελ. Ευχαριστώ. Θερμά τον εισηγητή για την ε, έκθεση αυτή των 80 σελίδων για ένα θέμα που αφορά 4.000 θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεστε κάνοντας πολύ συγκεκριμένες κατηγοριοποίησεις στην έκθεσή σας στις διάφορες εγκαταστάσεις που αφορούν ε, τουριστικές ε, εγκαταστάσεις, ψυχαγωγίας, μεταφορά προσώπων, ε, προϊόντων και πραγματικά, αν συγκρίνει κανείς αυτά που προτείνεται με όλα αυτά τα οποία έχουν ξεκινήσει πραγματικά στην Επιτροπή και σε άλλους ε, οργανισμούς, θα σας πω ότι πραγματικά και ειλικρινά εκπλήσωμαι για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά γίνονται αυτές οι εργασίες παράλληλα θα έλεγα. Σκέφτομαι βεβαίως ότι είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα και ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια τεράστια εργασία για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο και μικρό τομέα, ο οποίος αφορά πολύ λίγες δραστηριότητες. So, the commission Η Κομισιόν ε, θέλει να σχολιάσει. Είναι εδώ ο Λουίς Φιλίππε Γκεράρ. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ. Να προσπαθήσω να διευκρινίσω κάποια πράγματα, διότι ρώτησε κάποιος γιατί αναφερόμαστε σε δεν έχουμε μάλλον στο πεδίο εφαρμογή ε, κινητό εξοπλισμό ε, για ε, γιορτές και μηχανήματα σε πανηγύρια και Λούνα Πάρκ. γιατί μας αφορά καθαρά η μεταφορά ατόμων, δεν θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή σε κάτι άλλο, θέλουμε να μείνουμε σε αυτά. Όσον αφορά τα ιστορικά σειρματόσκηνα, αυτά εξαιρούνται, αφήνονται στην εθνική νομοθεσία και ε, ελπίζουμε ότι ο ορισμός των ιστορικών αυτών ε, εγκαταστάσεων ε, θα βρει σύμφωνες στις χώρες μέλη. Τώρα, όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, τι ακριβώς έχει γίνει με τις προτινόμενες τροπολογίες, περιλαμβάνεται το κεφάλαιο που περιλαμβάνεται και στο NLF, στο New Legal Framework και εμείς θεωρούμε ότι το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και για τον προσωπικό ε, εξοπλισμό προστασίας και τις συσκευές αερίου και μόλις ε, ε, εγκριθεί ο κανονισμός για την εποπτεία της αγοράς από την Επιτροπή οι διατάξεις αυτές θα αντικαταστήσουν αυτό που έχουμε στην τομεακή νομοθεσία για την εποπτεία της αγοράς που σημαίνει ότι Ό,τι έχουμε στη δέσμη μέτρο του ΕΝΕΛΕΦ και αυτό που θα έχουμε σε αυτόν τον κανονισμό ε, που συζητάτε τώρα για θέματα εποπτείας της αγοράς θα αντικατασταθούν από τον κανονισμό. Αυτό ε, θεωρούμε εμείς. Όσον αφορά την έκθεση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τις τροπολογίες που προτείνονται. θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν τον προτινόμενο κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Thank you. Um, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα. πέρα από τις άλλες τρεις εκθέσεις που αφορούν το θέμα της εποπτείας αγοράς και πέρα από το γεγονός ότι έχω την εντύπωση ο τριμερής διάλογος για τις τρεις αυτές εκθέσεις που αφορούν αυτό το πακέτο θα γίνει ταυτόχρονα, θα ήταν καλό να υπάρξουν συναντήσεις ε, μεταξύ των εισηγητών των τριών αυτών εκθέσεων περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας γι' αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και το θέμα της εποπτείας της αγοράς, καλό θα ήταν να υπάρξει ταυτόχρονα τιμερής διάλογος. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Έχετε το λόγο. Uh, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις διάφορες πολιτικές ομάδες για την υποστήριξη ε, όσον αφορά την έκθεση και για τις τροπολογίες. Το θέμα των ιστορικών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη βεβαίως ε, που αναφέρθηκαν σε αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν και κάποιες νέες εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει θέμα ασφάλειας. Το θέμα είναι η ασφάλεια. Αναφερόμαστε σε εγκαταστάσεις με σειρματόσχηνα και ο παράγοντας ασφάλεια είναι, αν θέλετε, το σημείο κλειδί. Και βεβαίως μπορώ να ενσωματώσω όλες σας τις προτάσεις Κοίταξα τις τροπολογίες και φυσικά και θα ενσωματώσω όλα αυτά που προτείνετε, τα οποία θεωρώ εξάλλου ότι ακολουθούν την ίδια γραμμή. Το θέμα των τουριστικών εγκαταστάσεων τώρα. Στην ε, Μαγιόρκα που είναι στην εκλογική μου επικράτεια το θέμα του τουρισμού είναι ένα μείζον θέμα. Γνωρίζω λοιπόν τα θέματα αυτά, τις επιπτώσεις του και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ναι, βεβαίως ε, είπατε ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις που αφορούν 4.000 θέσεις απασχόλησης, όμως εάν συμπεριλάβουμε τον τουριστικό τομέα τις τουριστικές εγκαταστάσεις καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για τεράστιες θέσεις, τεράστιο αριθμό θέσεων απασχολής και βεβαίως οι επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικές. Προσπάθησα λοιπόν να ενσωματώσω και αυτόν τον τομέα στην έκθεσή μου Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη που εκφράσατε. Φυσικά και χρειάζεται μετάφραση για να μπορέσει κανείς να εξετάσει προσεκτικά το κείμενο αυτό. Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος στο θέμα αυτό, είμαι Ισπανός και φυσικά και χρειάζεται χρόνος και θα περιμένουμε όλα τα κείμενα ε, να τα πάρετε ο καθένας στη γλώσσα του. Ευχαριστώ. Να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο να αλλάξουμε την ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών. Ε, να την μεταφέρουμε μετά τα Χριστούγεννα, εντάξει. Την πρώτη μέρα μετά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές. Το επόμενο σημείο στην ημέρη σε διάταξη. By the Commission of the Impact Assessment είναι η παρουσίαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής της αξιολόγησης επιπτώσεων για το θέμα της ε, αποκάλυψης εμπορικών μυστικών ε, και εμπορικού απορρίτου. Ε, κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψης αυτών των πληροφοριών. Να ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μήπως μπορείτε να βάλετε τις διαφάνειες ε, να φαίνονται πλήρως στην οθόνη. Επειδή έχω πολλές διαφάνειες, ε, να περάσω απευθεία στην παρουσίαση. Αυτό έρχεται σε απάντηση μιας συζήτησης που έγινε εδώ στην Επιτροπή μα ζητήθηκε να παρουσιάσουμε την αξιολόγηση των επιπτώσεων που έγινε για την πρόταση αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλέ διαφάνειες, ελπίζω να σας δοθούν και θα προσπαθήσω εγώ να τις διατρέξω κυρία Πρόεδρε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση στη συνέχεια. Να περάσουμε στην πρώτη ε, διαφάνεια είναι διαθέσιμες ε, διαδικτυακά και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, επομένως ε, μπορούμε να τις έχουμε. Να περάσω λοιπόν στην πρώτη ε, διαφάνεια και κατά πάσα πιθανότητα ίσως να καταφέρουμε κάποια στιγμή να τη συντονίσουμε. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω πάρα πολύ. Η γνώση βεβαίως είναι στο επίκεντρο της σύγχρονης οικονομίας και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας εξαρτάται από τις γνώσεις που καταφέρουν ε, να διαχειριστούν και να διαθέτουν. Και το όλο ζήτημα είναι ε, πώς ε, μπορεί κάποιος να αποκτήσει ιδιοκτησία της καινοτομίας. Μπορεί να γίνει και μέσω πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά κυρίως υπάρχει το θέμα της, του απορρίτου. Στην επόμενη διαφάνεια πιο συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση έχει κάποιες εμπιστευτικέ, πολύτιμες πληροφορίες στη διάθεσή της. Αυτές είναι αποδεικτικά στοιχεία και το άλλο στοιχείο είναι ότι τα εμπορικά μυστικά πάντα κάπου εμπλέκονται στην αλυσίδα. Για να σας δώσω μια εικόνα, πριν κάποιος ε, ε, λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για κάποια ε, εφεύρεση ή οτιδήποτε άλλο είναι εμπορικό απόρριτο και τα πάντα ε, βασίζονται στην αποκάλυψη αυτού του εμπορικού απορρίτου. Το εμπορικό απόρριτο λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο της ανταγωνιστικής οικονομίας και φυσικά της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στην επόμενη διαφάνεια. A key point. Can we have the next slide? I apologize. A key point ένα βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, ελπίζω κάποια στιγμή να βγει και η διαφάνεια, είναι ότι τα εμπορικά μυστικά δεν δίνουν στον κάτοχο κανένα δικαίωμα για τις πληροφορίες που δεν αποκαλύπτει. Δεν πρόκειται περί αποκλειστικού δικαιώματος εδώ μπορεί κάποιος ανταγωνιστής να ε, ανακαλύψει με νόμιμο τρόπο ακριβώς ε, ε, το ίδιο πράγμα και να καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι εργαλείο ανταγωνισμού αυτά τα πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο προχωρά κάποιος είναι με τον να συνεχώ συνεχώς και επομένως υπάρχουν επιπλέον εμπορικά μυστικά τα οποία έρχονται να προσθεθούν σε αυτά τα οποία διαθέτουμε. Αφετέρου, ένα βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτά τα εμπορικά μυστικά μπορούν να αποκτηθούν και παρανόμως, είτε μέσω κλοπής, είτε μέσω ε, κατάχρησης ή ίσως μέσω παραβίασης της εμπιστευτικότητας όταν μιλήσει κάποιος με έναν ε, ανταγωνιστή εταίρο. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα για να σας εξηγήσουμε λίγο τι κάναμε, προκειμένου να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση επιπτώσεων. Πρώτα, έγινε μια νομική μελέτη για να έχουμε μια γενική εικόνα της νομικής κατάστασης ε, στα 28 κρατημέλη. Στη συνέχεια έγινε μια πολύ καλή δημόσια ακρόαση, είχαμε μεγάλη συμμετοχή ε, και εκεί συζητήθηκε πώς θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε την αγορά και να λάβουμε πληροφορίες για το τι δεν διαθέτουμε αμέσως. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι οι επιχειρήσεις συνήθως δεν αποκαλύπτουν τα εμπορικά μυστικά τους. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα το οποίο μας απασχολούσε σε όλη αυτή την αξιολόγηση επιπτώσεων και ε, πιστεύω ότι το ερευνητικό τμήμα του Κοινοβουλίου πολύ καλά το διέγνωσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλλέξουμε αξιόπιστα δεδομένα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τελικώς βασιστήκαμε σε έρευνες. Ε, έγινε και μία δημόσια διαβίλευση βεβαίως, αλλά θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι η έρευνα για τον κλάδο που κάναμε είχε επικεφαλή τον ε, καθηγητή Φραντσόνη, ο οποίο είναι εμπειρογνώμονα επί του θέματος ε, από το Πανεπιστήμιο τη Μπολόνιας και ε, τήρησε τα όσα προβλέπονται στο μνημόνιο του Όσλο για τη μεθοδολογία. Επομένω, είναι ένα από του βασικού εκπροσώπους ε, στα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείτε ότι το 60% του δείγματο μας ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι στο οποίο θα επανέλθω αργότερα. Γίνονται φυσικά και δημόσιες ε, έρευνες, δημόσιες διαβουλεύσεις και θα δείτε ότι είχαμε περίπου 386 απαντήσεις ε, και αυτές όλες ε, ήταν σε διάφορες κατηγορίες φυσικά για να καλύψουμε όλο το ε, 152 ε, πολίτες ε, απάντηση βέβαια που έλαβε το κοινοβούλιο δεν είναι και πάρα πολύ μεγά, πολλές απαντήσεις αλλά ε, είχαμε πολλές απαντήσεις από επιχειρήσεις κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει επίσης το θέμα της ε, στάθμισης είχαμε μία απάντηση από την ε, Business Europe που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη και μία απάντηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μας δίνει την ίδια ε, στάθμιση. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα σε όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Ένα ακόμα θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω όσον αφορά τις απαντήσεις των πολιτών αφορά το γεγονός ότι περίπου οι μισές απαντήσεις ήταν ακριβώς οι ίδιες. Παρακολούθησα το έντυπο το οποίο είχε δοθεί ε, στο διαδίκτυο από κάποια πολιτική ομάδα, από κάποιο πολιτικό κόμμα, το οποίο ναι, είναι αποδεκτό, αλλά ε, αυτό το λάβαμε υπόψη μας στην εκτίμηση επιπτώσεων. Δεν μπορούμε να λάβουμε θέση από αυτό, αλλά μπορεί και να συμβεί. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν. Έχει 25 παραρτήματα νομίζω η εκτίμηση επιπτώσεων και καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να σας τα αναλύσω όλα εδώ. Ε, στην εκτίμηση, στη διαφάνεια αυτή έχουμε τα βασικές μας διαπιστώσεις. Καταρχάς το εμπορικό απόρριτο, τα εμπορικά ε, μυστικά όπως σας είπα είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, το θέμα της ε, ε λανθασμένης χρήσης, ε, της απόκτησης παρανόμως αυτών των εμπορικών μυστικών είναι ένα πρόβλημα. Και τρίτον, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό για την Επιτροπή σας, ε, διαπιστώσαμε ότι σίγουρα υπάρχει ένα κατακαιρματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, θέματα αντιμετώπισης της παράνομης απόκτηση εμπορικών μυστικών. Και αυτό φυσικά είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο το οποίο ε, μας ενδιαφέρει. Επόμενο θέμα είναι ποιε είναι οι συνέπειες του γεγονότος αυτού. Ε, εμείς πιστεύουμε και νομίζω ότι αυτό ε, το δείχνει και η έρευνα ότι υποσκάπτει την ε, διασυνοριακή καινοτομία και αυτό που κάνουν οι επιχειρήσει τη σήμερα ημέρα είναι να εξειδικεύονται σε συγκεκριμένου τομεί και να συνεργάζονται διεθνώ με εταίρου για να μπορέσουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα και αυτό ο κατακαιρματισμό προφανώ έχει ε, αρνητικέ συνέπειε. Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την αναζήτηση εταίρων αλλού στην ευρωπαϊκή αγορά και αυτό φυσικά ε, υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα στην εσωτερική αγορά εν γέννη. Όσον αφορά τώρα την οικονομική απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να δείτε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά και για τις μεγάλες αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα δείτε και από κάποια στοιχεία αργότερα ε, και στα όσα περιλαμβάνονται και στην εκτίμηση επιπτώσεων ότι υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη για την πρόταση αυτή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι επιπλέον το οποίο θα ήθελα να τονίσω σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι τα εμπορικά μυστικά διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία ε, ανταλλαγής ε, πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της καινοτομίας. Η ε, συνεργασία στην έρευνα είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικά στοιχεία και επομένως ε, αυτό είναι σημαντικό και για τα πανεπιστήμια και για εμπορικές επιχειρήσεις ε, και κυρίως για τα πανεπιστήμια που αναζητούν ε, εταίρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα όσα βρίσκουν στις έρευνές τους. Επομένως και αυτό σημαντικό στοιχείο για την εσωτερική αγορά. Τώρα, παράνομη απόκτηση. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι και τι διαπιστώνουμε εδώ. Σαφώς υπάρχει οικονομία της γνώσης, επομένως οι πληροφορίες είναι στο επίκεντρο κάθε επιχείρησης και υπάρχει μεγαλύτερη χρήση ε, φυσικά και ε, ε, βασίζονται όλοι στο απόρριτο. Από εκεί και πέρα, εξωτερική ανάθεση, αδειοδότηση, ένα σωρό άλλα στοιχεία αυξάνονται συνεχώς και αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται διαφορετικά οι ανταγωνιστικέ επιχειρήσει, δημιουργούν δίκτυο και επομένω ε, ο κίνδυνος διαρροή ε, πληροφοριών είναι ακόμα μεγαλύτερος. Ε, εξειδικευμένοι εργαζόμενοι αυξάνονται επίσης και αυτό σημαίνει ότι μετακινούνται και αυτοί εκτό των συνόρων και αυτό φυσικά θα μπορούσε να βοηθήσει και ένα βασικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει μικρότερο κύκλο παραγωγή. Ε, πολλές αναφερόμαστε σε προστασία και πολλά προϊόντα ε, μπορεί να έχουν χρόνο ζωής που να μετρέται σε μήνες. Δηλαδή ε, το θέμα είναι να μην διαδοθεί το εμπορικό μισθοκίκο και να μπορέσει κάποιος να εργαστεί με βάση αυτό. Και υπάρχει τώρα και το νέο που δεν είναι πια νέο, ε, το διαδίκτυο που το έχουμε εδώ και 20 χρόνια, τα πάντα γίνονται διαδικτυακά και φυσικά το hacking ε, ε, εδώ χρησιμοποιείται πολλές φορές για παράνομη απόκτηση εμπορικών μυστικών όπως σας είπα και νωρίτερα, τα δεδομένα πάντα αποτελούν πρόβλημα. Το να γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά τι γίνεται είναι πολύ σημαντικό. Ε, αναφέρθηκα στην έρευνα που έγινε για το ε, κλάδο που είναι η έρευνα που έχει και το πιο ανταποπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων και θα δείτε ότι οι επιχειρήσεις ήταν διατεθειμένες να μας πούν ότι είχαν υποστεί τέτοια παράνομη απόκτηση εμπορικών ε, ε, και επιχειρηματικών πληροφοριών και αυτό ήταν εις βάρος τους φυσικά ε, γιατί έχει πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες, όχι μόνο για την απόδοση των επιχειρήσεων, αλλά και για τα ε, στιμές των μετοχών όταν πρόκειται περί μεγάλων επιχειρήσεων. Ε, Υπάρχουν κάποια παραδείγματα, ακόμα και αυτή την εβδομάδα για παράδειγμα, μαθεύτηκε ότι υπήρξε ε, μια πολύ μεγάλη ε, αποκάλυψη πληροφοριών σε μια επιχείρηση ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες και ε, έγινε επίθεση από hackers και δόθηκαν στοιχεία, έλαβαν στοιχεία περίπου μια εβδομάδας, ακόμα και διάφορες εκδηλώσεις που είχαν οργανώσει. Εδώ έχετε μια διαφάνεια που σας δείχνει μια εικόνα για το πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα στα νομοθεσία των κρατών μελών με διάφορες ε, νομολογίες και ε, νομικά συστήματα. Πολλά ε, μέλη μπορεί να σκεφτούν ότι ορίστε υπάρχουν διαδικασίες αντιμετώπισης του φαινομένου, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικές οι δυνατότητες που προσφέρονται στα κράτη-μέλη και ακόμα και σε περιπτώσεις όπου καλύπτονται από την νομοθεσία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη νομικής ασφάλειας, ασφάλειας δικαίου σε αυτή την περίπτωση. Το ουσιαστικό εδώ, και να σας τονίσω κάποια στοιχεία, Δέκα κράτη-μέλη μόνο έχουν ορισμό του εμπορικού μυστικού των επιχειρηματικών πληροφοριών και ε, οι ορισμοί αυτοί, ε, παρά το γεγονός ότι καλύπτονται ήδη στις συμφωνίες TRIPS, ε, είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Υπάρχει επίσης και μεγάλη διαφορά ως προς τη δυνατότητα εκμετάλλευσης εμπορικού μυστικού από τρίτο δεν υπάρχει καμία αντιμετώπιση για χρήση από τρίτο ε, ενός μιας επιχειρηματικής πληροφορίας και υπάρχουν και έξι κράτη-μέλη που δεν έχουν συγκεκριμένη νομοθεσία επί του θέματος και βασίζονται σε γενικότερο αστικό δίκαιο. Που δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και τίποτα, αλλά αν κάποιο είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ακόμα και τα νομικά ε, στοιχεία, δεν ξέρει πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει και τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και στη διαφάνεια εδώ βλέπετε επίσης ότι υπάρχει έκκληση για προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο από πολλές επιχειρήσεις. Ένα ακόμα παράδειγμα εδώ, όσον αφορά το διορθωτικά μέτρα, Έχουμε κάποια διαγράμματα, τα οποία θα σας τα πω λίγο εντάχει, όσον αφορά την παραβίαση και τις διαδικασίες επί παραβάση ε, λόγω ε, Αποκάλυψη επιχειρηματικών πληροφοριών σε 7 κράτη-μέλη δεν υπάρχει καν δυνατότητα καταστροφής ε, ε, αγαθών. Ε, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κατακαιρματισμός. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, σαφώς υπάρχουν διαφορές και βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας το γεγονός ότι αυτές οι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών δεν μας επέτρεψε να κάνουμε αυτή τη διαμεθοριακή έρευνα στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτές τις διαμεθοριακές περιπτώσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αδύναμος ε, κρίκος είναι πάντα το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει προστασία στη χώρα σας, αλλά αν υπάρχει ένα δίκτυο επιχειρήσεων με το οποίο συνεργάζεστε ε, διεθνώς αν ένας από αυτούς βρίσκεται στην πιο αδύναμη περιοχή εκεί θα είναι και ε, το σημείο στο οποίο δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και να υπάρχει και κάποια ποινή. Όσον αφορά το βασικό ζήτημα το οποίο προέκυψε, ελοχεύει ένας κίνδυνος και μάλιστα είναι και υπαρκτός κίνδυνος όταν κάποιος προσπαθεί να επιλύσει μια διαφορά ε, αποκάλυψης πληροφοριών. Σε ορισμένες χώρες η απόπειρα να παραμείνει αυτό το εμπορικό μυστικό σε κάποιους κύκλους για να μπορέσει να υπάρξει δίκαιη δίκη δεν είναι πάντα δεδομένη. Ορισμένες φορές πρέπει να γίνει ανοιχτή ακρόαση και ακόμα και αν υπάρχει νομοθεσία δεν χρησιμοποιείται και ε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, αναφέρθηκα και στο ποινικό δίκαιο, Επικεντρώθηκα βέβαια στο αστικό δίκαιο, αλλά υπάρχει και ποινικό δίκαιο σε 12 κράτη-μέλη που επιβάλλουν κυρώσει επί του θέματος αυτού. Εδώ έχουμε την εικόνα. Τα... τα κενά είναι τα λευκά κουτάκια. Είναι ένας ακόμα τρόπος να δείτε πόσο κατακαιρματισμένη είναι η κατάσταση. Και τέλος, δεν είμαστε οι μόνοι που ε, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και ο ΣΑ ασχολείται με το θέμα. Εδώ έχετε ένα παράδειγμα και εξετάζει το επίπεδο προστασίας, ε, χρησιμοποιούν ε, οικονομικούς δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τον τομέα αυτό και τα τέσσερα μεγαλύτερα κράτη-μέλη έχουν πολύ μεγάλες διαφορές ε, αντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτά θα σας τα πω βιαστικά γιατί όπως σας είπα το πρόβλημα είναι ότι ελάχιστες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή υπερασπίζονται τι επιχειρηματικέ του πληροφορίες, κυρίως λόγω αυτού του κατακαιρματισμού και της έλλειψης σαφήνεια του νομικού συστήματος και από ό,τι βλέπετε το 29% αυτών που απάντησαν στην έρευνα είπαν ότι δεν υπάρχουν και αποτελεσματικά μέτρα και ένα 14% λέει ότι φοβούνται ότι θα χαθούν οι επιχειρηματικές τους πληροφορίες. Τα δύο λοιπόν βασικά προβλήματα τα οποία υπογραμμίσαμε σε αυτήν την ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων είναι ότι <clears throat> θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα και θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αποτροπής, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές τέτοιες ε, δραστηριότητες. Σημαντικά μειώνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό φέρεται ξεκάθαρα από την αξιολόγηση επιπτώσεων. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να μετρηθούν όλα αυτά, παρόλα αυτά αυτή είναι η γενικότερη τάση που διαπιστώσαμε. Κοιτώντας την πρώτη δυσκολία που σας παρουσίασα, είναι σαφέστατο ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτή η αβεβαιότητα οδηγάει τελικά σε μια πολύ ε, λιγότερη επιμονή όσον αφορά την καινοτομία και τις τεχνολογικές λύσεις. 40%, 40 των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμούν να μοιραστούν με άλλους, ε, να συνεργαστούν αν θέλετε, στον τομέα αυτό γιατί φοβούνται ακριβώς αυτήν την ε, υποκλοπή επαγγελματικών και εμπορικών ε, μυστικών. Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, 56% αυτών που συμμετείχαν μίλησαν για μείωση ανταγωνιστικότητας, ε, για απώλεια πελατών και συμβάσεων, συμβολέων. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι σαφέστατη η επίπτωση κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ε, σαφώς ε, εξαρτώνται και πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τέτοια κλοπή εμπορικών ε, μυστικών σε σχέση με τους μεγάλους πολιτικούς ομίλους. Υπάρχουν και κάποιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και από ό,τι φάνηκε από την μελέτη μας στα κράτη-μέλη που υπάρχει πολύ πιο αδύναμη προστασία φυσικά και η ανησυχία και ο κίνδυνος εμφανιζόταν πολύ υψηλότερος. Κάτι άλλο σημαντικό είναι αν θέλετε οι επιπτώσεις ε, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα στην αγορά απασχόλησης. 30 με 70 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης χάνονται εξαιτίας της βιομηχανικής κατασκοπίας και των επιπτώσεων της και αυτό είναι κάτι που δείχνει το εύρος του προβλήματος. Κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουν εδώ όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό είναι το θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων. Δηλαδή βλέπουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία όταν παρουσιάζει αδυναμίες δείχνει ότι η άμεση συνέπειες επί της ανταγωνιστικότητας και επί της ε, δυνατότητας ε, κινητικότητας των εργαζομένων είναι αλληλένδετες. Βλέπουμε δηλαδή ότι η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε κράτη-μέλη με χαμηλό επίπεδο προστασίας είναι διαφορετική. Υπάρχει δηλαδή μια αποτροπή, ένας αποτρεπτικός χαρακτήρας μιας υψηλής νομοθεσίας, μιας αυστηρής νομοθεσίας που προστατεύει ε, το εμπορικό και το επαγγελματικό απόρριτο. Η προστασία λοιπόν του εμπορικού αυτού απορρίτου και της καινοτομίας είναι κάτι που αναγνωρίζεται σαν πάρα πολύ σημαντικό από τις επιχειρήσεις. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν της ε, νομοθετικής προστασίας σε όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που διαφαίνεται από αυτήν την έρευνα και όπως είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου, φυσικά οι συμφωνίες, οι εμπορικές συμφωνίες TRIPS προβλέπουν πάντα μια τέτοια προστασία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης στην εσωτερική αγορά να διασφαλιστεί ομοιογένεια έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να είναι ανταγωνιστικές σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βεβαίως ένα θέμα νομοθετικής βάσης στην εσωτερική αγορά και το θέμα της ανάλυσης που κάναμε για την επικουρικότητα δείχνει ότι Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι οι χώρες που δέχτηκαν την αξιολόγησή μας όσον αφορά την πτυχή της επικουρικότητας. Τώρα, όσον αφορά τις λύσεις που προτείνουμε, τις εναλλακτικές λύσεις, βλέπετε εδώ ότι κάποιες από αυτές έχουν απορρευθεί. Ξεκινήσαμε με πέντε εναλλακτικές λύσεις, εναρμόνιση και φτάνουμε μέχρι τις ποινικέ κυρώσεις ενημέρωση βεβαίως και ευαισθητοποίηση, είναι το νούμερο 2. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει εδώ να επιλεγούν αυτές οι μη ρεαλιστικές λύσεις που βλέπετε ο κατακαιρματισμός ε, της αγοράς δεν μειώνεται οι συμφωνίες TRIPS ισχύουν εδώ και 20 χρόνια. Ο κατακαιρματισμός παρόλα αυτά δεν έχει μειωθεί και βλέπετε εδώ στην άλλη πλευρά αυτής της διαφάνειας ότι η γενική αντίδραση ήταν ότι χρειάζεται εδώ πραγματικά περισσότερη δράση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν ζητούν με σαφή τρόπο νομοθετική προστασία ή περισσότερη νομοθετική δραστηριότητα παρόλα αυτά ζητούν ε, κάποιες λύσεις και κάποια μέτρα. Βλέπετε εδώ την εναλλακτική λύση 5, εναρμόνιση αστικού και ποινικού κώδικα. Εμείς ε, θεωρούμε, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη της Επιτροπής, ότι η εναρμόνιση του ποινικού κώδικα βεβαίως είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το εξετάσει σαν την ίστατη λύση. Είναι πολύ νωρίς δηλαδή να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε θέματα όπως την κινητικότητα των εργαζομένων. Εξετάσαμε το θέμα αυτό στην μελέτη μας, αλλά βεβαίως θεωρούμε ότι δεν υπάρχει εδώ ε, αρκετή δυνατότητα για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια εναρμόνιση που θα πλήξει και την κινητικότητα των εργαζομένων. 7% λοιπόν βλέπετε των απαντήσεων ζητούν περισσότερη προστασία, 54% να μπορούν να ε, επιληθούν διαφορές και σε άλλα κράτη-μέλη, να γίνουν προσφυγές. Επίσης το θέμα του αποτρεπτικού χαρακτήρα μιας διαφορετικής νομοθετικής ενός διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει υποστήριξη, ε, ευρεία υποστήριξη μιας ε, περαιτέρω δραστηριοποίησης στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα, δεν χρειάζονται επεξηγήσεις. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους στοχεύσαμε το θέμα του ανταγωνισμού είναι στο επίκεντρο βεβαίως των, της ανησυχίας, το θέμα της νομικής αβεβαιότητας, το θέμα της ρήτρα για τις καταχρήσεις. Και βεβαίως το θέμα των ε, ενδυνάμει διαφορών που μπορεί να προκύψουν σε ένα άλλο κράτος μέλος και ε, η αυστηρότερη, η μεγαλύτερη προστασία η οποία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία νέων ε, εμπορικών εμποδίων και φραγμών. Αυτό είναι μια ανησυχία που ακούστηκε. Προσπαθούμε λοιπόν εδώ να καθησυχάσουμε αυτές, ε, αυτούς τους επιχειρηματίες που ανησυχούν για κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι κανόνες πιο σαφείς όσον αφορά την προστασία των εμπορικών, ε, του εμπορικού απορρίτου είναι κάτι που θα διευκολύνουν την ε, επιχειρηματική κοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας στην Επιτροπή προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ένα κείμενο με ισορροπία. Με σκοπό να διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ βεβαίως αναφερόμαστε σε εργαζόμενους ε, με κατάρτιση, με δεξιότητες συγκεκριμένες και βεβαίως χρειαζόμαστε και πολύ σημαντικές διασφαλιστικές δικλίδες. Γι' αυτό σας μίλησα για ισορροπημένο κείμενο το οποίο δεν θα παρεμποδίσει αυτήν την κινητικότητα των εργαζομένων. Το θέμα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης, των whistleblowing, της προστασίας τους και σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν θα πρέπει αυτή η προστασία του εμπορικού και επαγγελματικού απορρίτου να ε, δημιουργήσει περιορισμούς σε αυτήν την ελευθερία έκφρασης. Νομίζω ότι σας παρουσίασα την έκθεση στον τομέα αυτό, αλλά αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για όλα αυτά τα θέματα, με μεγάλη χαρά θα σας απαντήσω. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των συστάσεων της ενημέρωσης, πληροφόρησης, δεν θεωρούμε ότι ένα τέτοιο εργαλείο δαπανηρό θα βοηθήσει τη μείωση του κατακαιρματισμού και θα έχει θετικά αποτελέσματα όπως σας προανέφερα. Σας εξήγησα επίσης γιατί το θέμα της εναρμόνισης ε, του ποινικού κώδικα είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα όπως δημιουργία εμποδίων για την κινητικότητα των εργαζομένων, κάτι το οποίο θα ξεπεράσει τα ενδεχόμενα θετικά αποτελέσματα μιας τέτοιας προσπάθειας. Πρόεδρε, Νομίζω ότι τα υπόλοιπα δεν θα τα παρουσιάσω, αναφέρονται στις οδηγίες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ, είναι η τελευταία διαφάνεια στο σχέδιο αξιολόγησης Φυσικά και όλοι γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα νομικών μέτρων και νομοθετικών μέτρων δεν ε, διαπιστώνονται άμεσα, χρειάζεται χρόνος. Θεωρούμε λοιπόν εδώ ότι ακριβώς επειδή συνεργαζόμαστε με το παρατηρητήριο για τις ε, διαδικασίες επί και άλλους οργανισμούς που εξετάζουν τα δεδομένα και τους δείκτες και επειδή βεβαίως έχουμε ήδη ξεκινήσει μία εξέταση αυτών των δικτών, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένουμε έτσι ώστε η αξιολόγηση που θα γίνει να είναι η ε, ορθή, να βασίζεται σε σωστά στοιχεία είναι μια αξιολόγηση αντικτύπου και επιπτώσεων που πραγματικά συμπεριλαμβάνει πάρα πολλούς παράγοντες. Σίγουρα μακρηγόρησα, αλλά το θέμα ήταν τέτοιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Θα ήθελα τώρα να δώσω στην κυρία Κόμη την εισηγήτρια το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει και εγώ να πάρω λίγο χρόνο, διότι επειδή ήταν τόσο αναλυτική παρουσίαση, θεωρώ ότι θα πρέπει και εμείς τώρα να επισέλθουμε σε διάφορες λεπτομέρειες. Ε, σήμερα ε, συνεχίζουμε τη συζήτηση που ξεκίνησε σε προηγούμενη συνεδρίαση για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που θα ασχοληθεί, όπως είπαμε, με το εμπορικό απόρριτο. Να σας πω ότι εμείς εκφράζουμε μόνο γνωμοδότηση για τις πτυχές της εσωτερικής αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, επομένως και οι τροπολογίες μας θα είναι για τη γνωμοδότηση. Η Επιτροπή Ήτρεθα Αρμόδια Επιτροπή, η Επιτροπή Νομικών κοινωνικών Εγώ θεωρώ ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ω στόχο έχει να καθορίσει κάποιου κανόνε προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που καινοτομούν. Επειδή ακριβώ βιώνουμε κρίση, ό,τι μπορεί να βοηθήσει να ενισχύσουμε τον ε, βιομηχανικό ιστό μας, κυρίως τον ιστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξίζει την υποστήριξή μας. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο προσκήνιο για την επιστήμη και τις καινοτομίες και είναι ευπρόσδεκτο φυσικά και ένα σύστημα εναρμόνισης. Και είναι εύκολο να αντιλαφθεί κανείς πώς η δημιουργία νέων προϊόντων ή κάποιες καινοτόμες ιδέες ε, θα πρέπει να έχει κάποια ε, στοιχεία απορρίτου. Δυστυχώ, τα θέματα πνευματική ιδιοκτησία δεν καλύπτουν όλε τι περιπτώσει όσον αφορά τη δημιουργία κάποιου νέου ε, στοιχείου και τι πληροφορίε, οι οποίε θα πρέπει να είναι εμπιστευτικέ. Υπάρχουν πάρα πολλέ πληροφορίε που έχουν και οικονομική αξία και είναι θεμελιώδη σημασία για την ανταγωνιστικότητα των ιδεών τη επιχείρηση και διαφεύγουν πέρα από το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τα, ε, εμπιστευτικά, τα εμπορικό απόρριτο είναι ένα επιπλέον στοιχείο για την ε, μη τεχνολογική καινοτομία και προστασία. Επομένως θα πρέπει να βρούμε ένα καλό τρόπο για τη χρήση του εμπορικού απορρίτου. Θα ήθελα τώρα να περάσω σε κάποιες λεπτομέρειες, διότι αναλύοντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να έχουμε κατά νου το βασικό στόχο της οδηγίας, δηλαδή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Υπάρχουν διάφορα συμφέροντα και εγώ θα ήθελα το τελικό αποτέλεσμα να είναι η κατάλληλη ισορροπία ε, μεταξύ όλων των απόψεων. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες ε, σκέψεις φωναχτά, γιατί αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να ακούσω και τις προτάσεις και τις γνώμες όλων των συναδέλφων και φυσικά και τις πολιτικές τους θέσεις. Να περάσω στις λεπτομέρειες λοιπόν των όσων μόλις ακούσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δύο μελέτες, μία έρευνα και μία δημόσια διαβούλευση. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση Ήδη η Επιτροπή μας είπε ότι το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό ε, έχει άποψη για την βάση που αναλύθηκε. Έχουμε 386 επαφές, από τις οποίες 152 ε, ήταν ε, πολίτες και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο των επιχειρήσεων, διότι οι οργανώσεις όπως η Business Europe ή ε, οι οργανώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πολλές άλλες επιχειρήσεις εξέφρασαν την άποψή τους και επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια καλή βάση. Το πρόβλημά μου είναι για τους πολίτες, διότι 152 πολίτες είναι πολύ λίγοι. Ε, ως διαβούλευση θα μπορούσαμε να τους έχουμε και μόνο για την περιοχή της Λομβαρδίας. Ε, άμα πάω πόρτα-πόρτα θα βρω 152 ανθρώπους. Επομένως πρέπει να δούμε τι γίνεται γίνεται και με την πτυχή αυτή, διότι έχουμε και θέμα προστασία καταναλωτών εδώ. Σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, λοιπόν, με τους ε, ε, πολίτες και τις επιχειρήσεις εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις. Κάποιοι είναι αντίθετοι, οι πολίτες είναι αντίθετοι κατά, ε, σε μια νομοθεσία για τα θέματα αυτά, ενώ οι επιχειρήσεις είναι υπέρ. Εγώ πιστεύω ότι ο όρος μυστικό, απόρριτο, θα πρέπει στο μυαλό των πολιτών να δημιουργεί την εντύπωση της έλλειψης διαφάνειας ε, ε, και επομένως ορισμένες φορές είναι δύσκολο να ε, κάνει κάποιος μια συνέντευξη με ένα πολίτη χρησιμοποιώντας τον όρο μυστικός διότι του δίνει την εντύπωση ότι δεν γνωρίζει κάτι και αυτό ίσως μπορεί να κατευθύνει για την άποψή τους. Δεν αντιλαμβάνεται κανείς γιατί οι πολίτες δεν θα έπρεπε να δεχτούν ευνοϊκά μια νέα νομοθεσία. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν αυτό. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα για ποιο λόγο δόθηκαν αυτές οι απαντήσεις για να αντιληφθούμε την άποψή τους. Εγώ ζήτησα το όνομα της, ε, Ευρω... την άποψη συγγνώμη, Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών αλλά ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση. Είναι ε, πολύ κατακαιρματισμένες οι απόψεις που δόθηκαν στην ε, εκτίμηση επιπτώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σήμερα έκανε την παρουσίαση αυτή ε, δίνοντας μας πιο αναλυτικά στοιχεία. Υπάρχει και μια πολύ σαφή διαφάνεια διαφάνεια και φάνηκε ε, εκεί ότι τα κράτη-μέλη έχουν τελείω διαφορετική νομοθεσία σε θέματα προστασίας εμπορικού απορρίτου. Επομένω, η λύση είναι μέσω μια οδηγία να προσπαθήσουμε να έχουμε σύγκληση τη εθνική νομοθεσία, προσθέτοντα έτσι και κατάλληλη ασφάλεια δικαία. Θα ήθελα καταρχά να ξεκινήσω από τα διάφορα κεφάλαια, ξεκινώντα από την αρχή. Κεφάλαιο 1, άρθρο 1 και 2. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την άποψή μου, είναι αρκετά ισορροπημένη, αν και εγώ θα προτιμούσα μια πιο αυστηρή και περιοριστική γενική προσέγγιση, και εδώ θα ήθελα να κάνω μία πρώτη σκέψη για το πεδίο εφαρμογή. Το άρθρο 1 περιορίζει το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία σε απόκτηση, ε, διάδοση και χρήση ε, παρανόμως ε, εμπορικών πληροφοριών. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα και να πούμε ότι η εθνική νομοθεσία που προβλέπει προστασία θα πρέπει να παραμείνει. Και υπάρχει και το θέμα αυτό το οποίο ε, απασχολεί και το Συμβούλιο που ξεκίνησε τι εργασίε του πριν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχο τη οδηγία θα πρέπει να είναι να καθορίσει κάποια ελάχιστα πρότυπα προστασία, επομένω κάποια ελάχιστα επίπεδα προστασία του εμπορικού απορρίτου στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορεί να υπάρξει μια ελάχιστη εναρμόνιση. Βεβαίω τα κράτη που έχουν υψηλότερη προστασία καλώ την έχουν, αλλά θα πρέπει να καλέσουμε τι χώρε οι οποίε, όπω φάνηκε από τη διαφάνεια δεν έχουν καν κάποια ποινική πτυχή επί του ζητήματο να φροντίσουν να υπάρχει κατάλληλη προστασία. Αυτά θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν και κίνητρο για την εσωτερική αγορά. Να περάσω τώρα στους ορισμούς. Οι ορισμοί δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, ε, συνάδουν και με τη Συμφωνία TRIPS, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και κάποια αιτήματα για πιθανές προστίκες, πάντα στα πλαίσια του συστήματος TRIP, που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα πληρέστερο κείμενο. Άρθρα 3 και 4 τώρα, κεφάλαιο 2. Ε, εκεί καθορίζεται πότε η απόκτηση, η χρήση και η διάδοση είναι νόμιμη ή παράνομη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιλέγει να ε, βγαίνει αυτό με βάση την αρχή της ενοχής. Γίνεται λοιπόν αναφορά στην πρόθεση ε, είτε με δόλο είτε από εμέλεια. Και αυτό φυσικά θα μπορούσε ίσως ε, να μας οδηγήσει και σε μια αντικειμενική αξιολόγηση για να υπάρχει καλύτερη προστασία του εμπορικού απορρίτου. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας από αυτού, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Όσον αφορά τα μέτρα τώρα και επομένως κεφάλαιο 3 πλέον, μέτρα, προστασία και ε, ε κυρώσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο θέμα αυτό για το ο, όσα προτείνουν από πλευρά εσωτερική αγοράς και καταναλωτών, αλλά για τις πτυχές ακόμα και αυτές θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, όσον αφορά τα συμφέροντα ε, ε, που, και ε, που απασχολούν το θέμα αυτό. Αναφερόμαστε στα θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία του ατόμου, του καταναλωτή, του επαγγελματία, αλλά φυσικά και επιχειρήσει και νομικό καθεστώς. Οι αιτιολογικοί σκέψη 23 και 24 είναι αφιερωμένες στο σημείο αυτό και φυσικά η νομοθεσία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειώνει την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Ο σεβασμός της χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, καθαρό επίπεδο προστασίας Υποτίθεται ότι συζητάμε την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Χαίρομαι που ζητάτε την συνεισφορά των συναδέλφων, αλλά ε, θα ήθελα να έχει και χρόνο η Κάρθριν Στάιλερ για να συζητήσουμε την ε, ε, δική της την έκθεση. Δεν έχω πολύ. Δύο λεπτά και ακόμα. Δύο λεπτά ακόμα. Θα τα πω γρήγορα. Γιατί ήθελα να θίξω κάποια σημεία και να συνεχίσω. Ωραία, θα τα πω γρήγορα, μην ανησυχείτε. So, at the end. <laughs> λοιπόν, εν τέλει. Να, συγγνώμη, να τα πω καλύτερα Ιταλικά. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας, διότι υπάρχουν κάποια πολύ ευαίσθητα θέματα. Συγγνώμη αν άρχισα να κάνω αναλυτική παρουσίαση, γιατί εμείς συζητάμε εδώ την εκτίμηση επιπτώσεων, αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα ε, στα οποία δεν λάβαμε απαντήσεις από τους πολίτες. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα και δεν χρησιμοποίησα ε, χρόνο σε ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά σε ιταλικά πρότυπα, αλλά επειδή ε, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, θα ήθελα να επικεντρωθώ στις λεπτομέρειες και όχι σε γενικόλογα πράγματα. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Ο κύριος Μωρέτη. Όχι. Μέρους των σοσιαλιστών. Δεν είναι εδώ ο κύριος Μωρέτη. Η κυρία Μακλάκιν από το ECR. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την Επιτροπή που μας παρουσίασε λεπτομερό το όλο θέμα. Χαίρομαι ότι γίνεται αυτή η εκμήρυση επιπτώσεων και στο τέλος το τελικό πίνακα μας δείχνει πολλά πράγματα μας απασχολούν. Ελπίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να βρουν έναν τρόπο να μην υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως θα πρέπει στις ΜΜΕ να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης διότι ξέρουμε ότι οι θέματα προσφυγών δεν έχουν πάρα πολλά χρήματα να διαθέσουν και θα πρέπει πάντα το ε, εμπορικό απόρριτο να μπορούμε να τους το εγγυόμεθα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ε, προσφυγές έχουμε έξι χρόνια στη διάθεσή μας θα πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα σωστό τρόπο να ενεργήσουμε. Κάτι άλλο που με απασχολεί είναι το κόστος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κόστος για αυτόν που υφίσταται το πρόβλημα. Μπορείτε επίσης να μας πείτε ότι οι χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ένα τέτοιο σύστημα ε, δεν θα πρέπει να το αλλάξουν με την εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. η κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ. Δεδομένου ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε αυτή την εκτίμηση επιπτώσεων και δεν έχουμε ακόμη δει το σχέδιο έκθεσης, έχοντας ακούσει τι είπε η συγγήτρια, θα ήθελα να κάνω την εξής γενική παρατήρηση. Αυτό με απασχολεί. Η εκτίμηση αντικτύπου βασίζεται στο ότι το θέμα της προστασίας του εμπορικού απορρίτου βασίζεται μόνο σε θέματα καινοτόμων επιχειρήσεων. Μήπως αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Τι εννοώ. Ότι η καινοτομία μεταξύ των επιχειρήσεων είναι το κύριο θέμα. Στην εκτίμηση όμως γίνεται λόγος γιατί ότι θα μας προστατεύσει η κοινοτική νομοθεσία από το πόδι. Τι θα γίνει όμως όταν υπάρχει συνεργασία μέσω ανοιχτών πηγών μεταξύ των επιχειρήσεων. Πώς μπορεί ο καθένας να προστατεύσει τα μυστικά που διαθέτει. Τώρα, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι όλα αυτά γίνονται υπέρ των ΜΜΕ. Αν δει κανείς την εκτίμηση επιπτώσεων και όπως είδαμε και σε μία από τις διαφάνειες, 125 εταιρείε απήντησαν, 59 από τις οποίες είναι μικρομεσαίες. Άρα όντως, όπως λέει η εκτίμηση ε, αντικτύπων, τα ωφέλη θα είναι μεγαλύτερα για τις μημία δεδομένου ότι δεν έχουν ε, τα οικονομικά μέσα να προσφύγουν να ζητήσουν νομική προστασία με την κοινοτική μονομοθεσία μήπως και πάλι δεν θα μπορούν οι ΜΜΕ να προσφεύγουν ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν αυτή την ε, δυνατότητα. Μήπως έτσι δυσχεραίνουμε την κατάσταση ακόμη περισσότερο για τις ΜΜΕ. Έχει γίνει περαιτέρω έρευνα ώστε να υπάρχει προστασία για αυτές. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής. Εργάστηκα ως δικηγόρος για 14 χρόνια και έχω πείρα επί του θέματος και είδα σε μία από τις ε, διαφάνειές σας ότι το εμπορικό μυστικό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και κάποιος άλλος ε, το εμπορικό πόρυτο να κάνει το ίδιο με σας. Πώς μπορείτε εσείς να εξασφαλίσετε το ότι αυτό το οποίο εσείς ε, παρουσιάζετε στην αγορά στα πλαίσια του εμπορικού απορρίτου είναι δικό σας. Πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι αν έχει κλαπεί από σας το εμπορικό απόρριτο έχετε υποστεί μια ζημία. Και πολλές φορές πολλοί λέγουν ότι αν δεν μου είχε κάποιος ε, κλέψει τις ιδέες μου ή το εμπερικό μυστικό θα είχα μπορέσει να έχω πολύ περισσότερα οικονομικά ωφέλη. Και σε τέτοιες περιπτώσεις η απάντηση συνήθως είναι ότι δεν έχουμε μέσα να το πολεμήσουμε αυτό το θέμα. Οι μεγάλη εμπορικοί επίσης εταίροι έχουν, ακολουθούν μια σχετική νομοθεσία όσον αφορά την παράνομη χρήση δεδομένων ή τεχνογνωσίες. Επίσης, τι έχουμε να κάνουμε με τις περιπτώσεις ε, κρατών όχι πλέον από οι Σοβιετικές, αλλά η Κίνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να μην επαναλάβω ότι είπα την τελευταία φορά για τον εκπληκτικό κάπως ε, τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εργασία αυτή. Νομίζω ότι ξεκινάμε από το τέλος και κατά την άποψή μου ο στόχος μας είναι πολύ μακριά από αυτόν που μας παρουσιάζεται. Πατάμε κουμπάκια Πρώτα απ' όλα τα ανταστοιχονομιστικά στην Ευρώπη. Βεβαίω, συμφωνούμε. Δεύτερον, η πράσπιση των συμφερόντων των ΜΜΕ. Προφανέ. Τρίτο, θα δημιουργήσουμε θέσει επασχόληση. Τέταρτο κουμπάκι. Όλα αυτά θα είναι θαυμάσια για την έρευνα και έτσι η Ευρώπη θα γίνει για θέματα απασχόληση κτλ. τα το πιο υπέροχο μέρο στον κόσμο. Δυσπιστώ εγώ πολλέ φορέ αυτά που ελέγονται για τις μιμίες. Στη Γαλλία τουλάχιστον οι εργοδότες των ε, μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων προασπίζουν το εμπορικό απόρριτο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν θα επαναλάβω αυτό το οποίο έλεγε. Αν δει κανεί 150 επιχειρήσει από εδώ και από εκεί και του ρωτήσει αν εμεί ε, εξασφαλίσουμε και οριστεύουμε το εμπορικό απόρριτο, συμφωνείτε, όλοι ναι θα πούνε. Αλλά εμένα πολλά πράγματα με απασχολούν με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα αυτό και για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα και την τελευταία φορά, θεωρώ ότι ο πίνακας αυτός μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Και όσον αφορά τη γαλλική νομοθεσία, την οποία γνωρίζω, διότι είμαι δικηγόρος για 25 χρόνια, φυσικό είναι, διότι είμαι πιο μεγάλη στην ελληνική από την κυρία Κάλλας, είναι η εξή. Στη Γαλλία το εμπορικό απόρριτο όταν είναι νόμιμο, διότι τι όρος δεν υπάρχει στην οδηγία και εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια νόμιμα συμφέροντα προσπιζόμαστε. Το δικό μας από νομικής πλευράς, ε, από αστικής πλευράς και από την ΚΝΑΟ προστατεύεται. Και αυτό γίνεται σε πολλές χώρες. Πάντα λοιπόν εγώ ήμουν δύσπιστος σε θέση με τα επιχειρήματα και τις διακηρύξεις που γίνονται με αυταχικό τρόπο. Ακούστε, σε κάθε χώρα υπάρχει νομοθεσία διαφορετική, σε κάθε χώρα το ξέρουμε, αλλά πολλές φορές μας λέγουν ότι πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα το αστικό και το ποινικό κώδικα και δεν λειτουργούν τον ίδιο τρόπο. Και τώρα μου λέγουν ότι Υπάρχουν διάφορα δελτία τα οποία παραβιάστηκαν και υπάρχουν διαδικασίες που έχουν ε, ε, παραβιαστεί ακόμα και στη ΣΥΠ. Ακούστε. Πρόκειται περί κλοπής. Μη μου λέτε λοιπόν ότι πρόκειται πάντα για εμπορικό απόρριτο θέλω να προσοδέψω. Υπάρχει το αστικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο, το οποίο προστατεύει την κλοπή. Σε ποιο μέτρο λοιπόν ένα εμπορικό απόρριτο που δεν ε, καθορίζεται και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στους καταναλωτές θα εφαρμοστεί. Τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Πώς ε, ξέρουμε ότι οι διάφορες ε, πολυεθνικές δεν θα πάνε στη ΣΥΠΑ και στα πλαίσια του TTIP δεν θα πούν ότι είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για όλες, σε όλους τους τομείς τους εμπορικούς. Και όλα, ό, όλα ό,τι γίνονται, γίνονται για να προστατευτούν οι καταναλωτέ που θα ξέρουν περί τίνο πρόκειται. Πιστεύω ότι η τη παρούσε κατάσταση είναι πολύ ε, ευρέω περιεχομένου και γενικού η οδηγία αυτή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Εμένα δεν μου απέδειξε κανεί μέχρι τώρα ότι όντω υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με την προστασία παραγωγής των TTIP ε, και των ΜΜΕ. Ευχαριστώ. Α, εκ μέρους της Γκουε, η Μαστάλκα δεν είναι εδώ. Από την EFD δεν έχει οριστεί ε, σκιώδης Ακόμη θα δώσω το λόγο σε μία συνάδελφο και μετά στην ε, κυρία, ακόμη και στην Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αυτό που μας απασχολεί είναι στα πλαίσια της εκτίμησης αντικτύπου αυτό που λέει η Επιτροπή ότι έτσι όπως προτείνει Τίνεται η οδηγία θα έχει ε, θετικές επιπτώσεις στην κινητικότητα των εργατικών χερών. Η τεχνογνωσία ενός εργαζομένου σε μια επιχείρηση νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα όταν κάποιος θέλει να βρει μια νέα δουλειά και κάποιος ο οποίος θέλει να προσλάβει ένα νέο εργαζόμενο κοιτάει στο, ε, τα προσόντα του και την ε, πείρα του και βεβαίω φέρει μαζί του κάθε νέο εργαζόμενο σε μια επιχείρηση όλη την τεχνογνωσία που διαθέτει από την προηγούμενη δουλειά στην οποία ήταν. Αν λοιπόν τα πάντα θεωρούνται εμπορικό απόρριτο χωρίς να υπάρχουν ε, ε, εξειδικεύσεις, πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να πάει σε μια νέα δουλειά και να προστατεύεται από το ότι κάποιος ενδεχομένως θα του πει ότι ε, μεταφέρει πληροφορίες που έπρεπε να κρατήσει μυστικές στα πλαίσια του εμπορικού απορρίτου και πώς μπορεί να το παρουσιάσει αυτό ένα από τα προσόντα που διαθέτει την πείρα του δηλαδή για τη νέα του δουλειά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ήμουν πολύ προσεκτική στην παρουσίαση που έγινε και στη συζήτηση που ακολούθησε, αλλά πραγματικά ανησυχώ γιατί πρώτον οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι όμιλοι μπορεί να ε, θεωρήσουν ότι ένα απόρριτο, ένα εμπορικό, βιομηχανικό, μυστικό μπορεί και πρέπει να προστατευτεί. Τι κάνουν όμως στην πράξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το αποκτήσουν αλλά και να το προστατεύσουν. Αξιότιμε συνάδελφοι από την Επιτροπή. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ περίεργα αυτά που μας λέτε. Οι διαδικασίες που προτείνετε καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολες, βαριές, χρονοβόρες, 8 χρόνια μας λέτε. Μα πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να αντέξει. Και εδώ υπάρχουν πολύ συχνά διαφορές που εμπλέκουν και τους εργαζόμενους και τους ε, εργοδότες, ποιος έκλεψε από ποιον, παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν τριμερείς θα έλεγα διαφορές πολλές φορές. Είναι βεβαίως ε, η νομοθεσία υπέρ συχνά του εργαζόμενου, τουλάχιστον στη Ρουμανία έτσι γίνεται. Και βλέπουμε ότι αν υπάρχει διαμάχη μεταξύ μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης και ενός μεγάλου ομίλου, μια μεγάλης επιχείρησης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει η μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι μόνο και μόνο το κόστος και ο χρόνος μιας τέτοιας διαδικασίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, το αντέξει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν πολύ πιο ε, συγκεκριμένα να συζητήσουμε τους ορισμούς, διότι κατανοείται κάτι τελείως διαφορετικό από μας ε, πίσω από τις λέξεις που χρησιμοποίησε. Το θέμα, παραδείγματο χάρη, των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα βοηθήσουμε και θα προστατεύσουμε με μια τέτοια οδηγία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν βλέπω τίποτα, ούτε στη μελέτη σας, ούτε σε αυτά που μας παρουσιάσετε. Τι να σας πω, ίσως δεν είχαμε αρκετό χρόνο, αλλά δεν καταλαβαίνω. Και ακούγοντας ε, την παρουσίαση της εισηγήτριας και ακούγοντας αυτό που λέτε εσείς από την Επιτροπή, μιλάτε για τη Συμφωνία TRIPS, αναφέρεστε στα μέχρι τώρα μέτρα, αλλά πραγματικά πώς μπορεί κανείς να αποδείξει ότι κάτι είναι εμπορικό ή επαγγελματικό απόρριτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο ορισμός και πραγματικά επαναλαμβάνω το αρχικό μου ερώτημα πώς θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ πάω στη χώρα μου πίσω και εξηγώ στους επιχειρηματίες στο μεγάλο δίκτυο των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ότι θα σας προστατεύσουμε. Πώς, δώστε μου επιχειρήματα. Θέλετε να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει, αλλά βεβαίως ε, μπορώ να απαντήσω και ειδικά σε κάποιες ερωτήσεις των ε, ε, αξιότιμων βουλευτών. Όσον αφορά τις ΜΜΕ, προσπαθούμε να έχουμε όσο πιο αντιπροσωπευτικό αριθμό μιμιέ μπορούμε και βασιζόμαστε σε διάφορες τεχνικές μελέτες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μιμιέ που έχουν πρόβλημα με αυτά τα θέματα και έχουμε εδώ μικρό αριθμό, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και ξέρω ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν ε, προβλήματα που ε, αναγνωρίζονται διεθνώς για το πρόβλημα που έχουν. Δεύτερον, πολλοί ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι οι ΜΜΕ δεν μπορούν εύκολα να προσφύγουν. Κάποιες το κάνουν. Δεύτερον, πολλές ΜΜΕ με τις οποίες μιλήσαν μας είπαν ότι το γεγονός ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι θα υπάρχουν κοινοί ορισμοί για κάποιες πρακτικές έτσι όπως το προβλέπουμε για την κοινωνική ε, για την κοινοτική νομοθεσία και ισοδυναμή με το TRIPS είναι κάτι το οποίο θα τις διευκολύνει διότι τελικά θα πρέπει να υπάρχει ε, μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Το ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί δημιουργεί πρόβλημα. Όντως λοιπόν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξει εναρμόνιση στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι όσον αφορά τώρα την ε, ε, η αξία του κειμένου αυτού για τις ΜΜΕ δεν θα πρέπει να το υποτιμάτε. Απ' την άλλη, δεν είναι μόνο θέμα προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περίπτωση διαφοράς. Πολλέ ΜΜΕ μα είπαν ότι αν πραγματικά έχετε ένα κοινό ορισμό και ένα σαφές κείμενο σχετικά θα βοηθηθούν όταν κάνουν κοινοπραξίες και συνεργάζονται με μεγάλες επιχειρήσεις. Διότι γνωρίζουν με σαφήνεια τι ακριβώς μπορούν να διαπραγματευτούν με αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Διότι υπάρχει τάσεις και κατανοώ πλήρως απόψεις των Ευρωβουλευτών ότι θα υπάρχουν λόμπι από τις μεγάλες εμπορικές εταιρείες των μεγάλων εμπορικών συμφερόντων. Αλλά ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρές μιμιέ. Και δεν είναι πάντα οι μικρές μιμιέ που μπορούν ε, να κατηγορηθούν ότι κάνουν κάτι το ανέντιμο. Και το αντίθετο συμβαίνει και θα πρέπει η κατάσταση να αποσαφινιστεί ώστε να έχουν περισσότερες δυνατότητες οι ΜΜΕ ε, διαπραγμάτευσης. Βεβαίως πάντα εντός περιορισμένων ορίων, αλλά εν πάση περιπτώσει από την άποψη των ΜΜΕ πιστεύουμε ότι εδώ υπάρχει προστιθέμενη αξία. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Ανέφερα στην παρουσίασή μου ότι με τον α ή β τρόπο, αυτό είναι κάτι που το προστατεύουν όλα τα κρατημέρη. Δεν είναι λοιπόν ε, θέμα ε, θέσει σε αμφισβήτηση τι γίνεται σε μία χώρα σχέση με την άλλη. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν διαφορές. Το επίπεδο προστασίας όταν βρίσκει κανείς σε μία διασυνοριακή περίπτωση συνεργασίας ή προβλήματος είναι ότι θα πρέπει να ξέρετε ε, από νομικής πλευράς ε, ποιοι κανόνες και νομοθεσία σας προστατεύει και πώς μπορείτε να προσφυγείτε. Και σήμερα το κόστος για αυτές τις μιμία είναι μεγάλο. Γι' αυτό τον ε, τρόπο κάποιες επιχειρήσεις δεν κάνουν κάτι τέτοιο, δεν προστέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Το είπαν πολλοί και παγώνουν τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ, λοιπόν, ε, όταν κάνετε λοιπόν μια πρόταση νομοθεσίας ή αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορούν οι ΜΜΕ να προσφεύγουν όταν ε, έχουν το δικαίωμα. Ξέρω από την πείρα μου τόσα χρόνια στην Επιτροπή ότι δεν τους αρέσουν αυτού του είδους οι, οι, διαδικασίες, αλλά εν πάση περιπτώσει όντως ε, εδώ βοηθούνται. Και πρέπει να σας πω ότι δεν γίνανε βιαστικά ότι έγιναν στα πλαίσια αυτή της ε, εκτίμησης αντικτύπου. Δεν θα το θέταμε επιτάπητο στο όλο θέμα αν ήταν στα τα πράγματα. Πιστεύω ότι προστατεύουμε τη σμήμια. Η συγγήτρια θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Ξέρουμε ότι για το θέμα αυτό θα συνεργαστεί με τους συναδέλφους σας να κάνετε μια καλή έκθεση. Θέλετε τώρα ολοκληρώνοντας να πείτε κάτι. Ναι, πολύ σύντομα. Αν δεν ήταν αυτό οδηγία υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που και εμείς θέλουμε να τις προστατεύσουμε ε, καλύτερα, δεν θα είχε και κανένα σκοπό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όσον αφορά τους χρόνους της δικαιοσύνης, ε, τι να σας πω, νομίζω ότι η Ιταλία συνεχώς είναι επιπαραβάση λόγω των μακρόχρονων διαδιοκοσιών και την ε, ε, ασάφεια των ποινών. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα το οποίο θα αντιμετωπιστεί στο θέμα αυτό. Χρειάζεται ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση. Εναρμόνιση του ευρωπαϊκού ε, συστήματος δικαιοσύνης. Αλλά αυτό είναι άλλο τομέα και αλλουνού αρμοδιότητα. Από τη δική μου την εμπειρία, γνωρίζοντας ε, στην Ιταλία την, εμπειρία, την κατάσταση όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, επικρατούν, πολλές φορές αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καινοτομούν. Εμείς δίνουμε χρηματοδότηση στις startups, στις νεοφυείς επιχειρήσεις για να καινοτομήσουν και αυτές είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να προστατεύονται διότι δημιουργούν μια νέα τεχνολογία που την χρησιμοποιεί στη συνέχεια η μεγάλη επιχείρηση. Ορισμένες φορές αυτές οι startup είναι ιδιοκτησίες μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ορισμένες φορές είναι είναι αυτόνομες και επομένως ε, συνεισφέρουν και θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός εναρμενισμένος ορισμός, να υπάρχει ένα ε, σημαντικό επίπεδο προστασίας και αν υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία σε κάθε κράτος μέλος, ευπρόσδεκτη. Εμένα η ιδέα μου ήταν να υπάρχει κανονισμός, είμαι υπέρ ποιων δραστικών μέτρων. Υπάρχει οδηγία και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο προκειμένου να προστατεύσουμε εργαζομένους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για την ε, πάρα πολύ αναλυτική παρουσίαση για την αξιολόγηση επιπτώσεων ε, και ε, θα το εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα. Επόμενο σημείο, έχουμε και πάλι παρουσίαση αξιολόγησης επιπτώσεων εδώ. Κυρία Τζιράου, θα παρουσιάσετε εσείς την αξιολόγηση επιστώσεων για τις συσκευές αερίου. Η Κάθριλ Σίλερ είναι η εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Και από ό,τι βλέπω είναι εδώ και η Άλισον Ντέιβις από το Τμήμα αξιολόγηση Επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα μπορέσει να παρεστεί σήμερα το απόγευμα. Αν έχουμε χρόνο λοιπόν και θέλετε να κάνετε σχόλια για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων ακόμα και για τα απογευματινά θέματα, ε, πολύ καλά. Αν έχουμε χρόνο θα τα συζητήσουμε ε, πρώτα αυτά. Ε, να δώσουμε όμως πρώτα το λόγο στην Επιτροπή, ο κύριος Ζηράου. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Βέζα Καταζήστο θα κάνει την παρουσίαση και μετά θα σχολιάσουμε. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Αν δούμε λοιπόν την πρώτη διαφάνεια. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο ε, στην παρουσίαση, αλλά θα ήθελα λίγο να σας παρουσιάσω την ίδια τη διαδικασία. Η οδηγία για τις συσκευές ε, αερίου είναι το ε, πλαίσιο για τις συσκευή αερίου και τις εγκαταστάσεις τους και υπάρχει από το 1990. Έχουμε λοιπόν μία ε, κλασική οδηγία νέου νομοθετικού πλαισίου η οποία ε, έχει καλά αποτελέσματα αλλά τώρα αναθεωρείται. Εποφεληθήκαμε και από την ύπαρξη μιας ομάδας εργασίας των κρατών μελών που υπήρχε ευθύ εξ αρχής από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή οδηγία και στα πλαίσια των συζητήσεων στην ομάδα εργασίας των κρατών μελών πολλά θέματα εντοπίστηκαν ε, στη διάρκεια των τελευταίων ετών η ομάδα εν τέλει ε, σύστησε μια ειδική task force για να συζητήσει ε, πιο διεξοδικά την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας και πέραν αυτού υπήρχε και μια εκ των υστέρων αξιολόγηση της κείμενης οδηγίας. Τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις και της Task Force και της Ομάδας Εργασίας ε, των Κρατών Μελών και του, ε, της αξιολόγησης εκ των υστέρων χρησιμοποιήθηκαν για να ξεκινήσει μια συγκεκριμένη μελέτη επιπτώσεων για τα διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και επιπλέον οργανώθηκε και μια δημόσια διαβίλευση προκειμένου να ρωτήσουμε τους ενδιαφερομένους κατασκευαστές, εργαστήρια, κοινοποιημένου φορείς, ε, ε, δημόσιες αρχές, πολίτες να μας πούν την άποψή τους και να μας κάνουν προτάσεις. Όλα αυτά συνεισέφεραν στην αξιολόγηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τελικώς οδήγησε στην έκθεση της εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία και εγκρίθηκε το Μάιο του 2014. Έχουμε τη νομική βάση και έχουμε και την έγκριση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Νομοθετική πρωτοβουλίας η οποία παρουσιάστηκε το Μάιο φέτος. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τρεις διαφορετικούς τομείς θεμάτων που πρέπει να εξετάσουμε. Ο πρώτος βεβαίως είναι πάντα η ευθυγράμμιση με, την, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια δέσμευση που ανέλαβαν τα θεσμικά όργανα και στην περίπτωση των συσκευών αερίου δεσμευτήκαμε προκειμένου να λάβουμε υπόψη όλες τις ε, οριζόντιες διατάξεις, τους ορισμούς και ούτε καθεξής που παρουσιάστηκαν και συμφωνήθηκαν στην απόφαση 768 του 2008. Αυτό σημαίνει ότι όπως και άλλες οδηγίες οι οποίες αναθεωρούνται και εμείς ε, λάβαμε υπόψη μας οριζόντιους ορισμούς, υποχρεώσεις οικονομικών φορέων, αξιολογήσεις συμμόρφωσης και τις διατάξεις για τους κοινοποιημένους φορείς και το καθεξής δεν ε, διαπιστώσαμε κάποιο σημαντικό πρόβλημα με τις οριζόντιες πτυχές ε, στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας για τις συσκευές αερίου, αλλά φυσικά υπήρχαν και κάποια θέματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Στην περίπτωση των συσκευών αερίου δεν υπήρχε όμως ανάγκη να πάμε, να πάμε πέραν της ε, ε, ευθυγράμμισης του νομικού κειμένου και επομένως οι αλλαγές οι οποίες ε, γίνονται δεν εισάγουν κάποια νέα στοιχεία στο νομικό πλαίσιο και οι συνέπειες είναι οι ίδιες ε, με τις υπόλοιπες εννέα οδηγίες που βρίσκονται σε αυτή τη δέσμη μέτρων του νέου νομοθετικού πλαισίου. Για να συνοψίσουμε ε, τι συνέπειες έχουμε. Πρώτον, δεν υπάρχει πολύ σημαντική συνέπεια στο κόστος για τις επιχειρήσεις και τους κοινοποιημένους φορείς. Η διαδικασία γίνεται κυρίως για να συμπληρέσουμε τις ε, ε, κείμενες υποχρεώσεις και να κωδικοποιήσουμε κάποιες πρακτικές οι οποίες ήδη εφαρμόζονται από τους ενδιαφερομένους του κλάδου. Επομένως, δεν υπήρχε δυνατότητα να υπάρξει κάποια ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων. Πρόκειται κυρίως ε, για ποιοτικά στοιχεία τα οποία απλώς ε, διαπιστώθηκαν και επίσης δεν υπάρχει κάποιο δυσανάλογο άκθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην όλη διαδικασία, αλλά Για παράδειγμα, το κόστος για τη δημόσια διοίκηση ε, μπορεί να ε, αυξηθεί λίγο, για παράδειγμα για γραπτή κοινοποίηση προς κοινοποιημένους φορείς. Τώρα, να περάσουμε στα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τον κλάδο. Μετά από την πολύ προσεκτική εξέταση όλων των συνεισφορών των ενδιαφερομένων, ε, εντοπίσαμε κάποιους τομείς ...στα οποίους θα έπρεπε να εξειδικεύσουμε στα πλαίσια της ε, αναθεώρησης. Πρώτο στοιχείο που έχουμε στη διαφάνεια, το να υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί για τον κλάδο στα νομικά κείμενα. Ένα από τα προβλήματα της ε, ε, η οδηγίες σε ενισχύ είναι παρά το γεγονός ότι υπάρχει ε, ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής ε, για διάφορες εφαρμογές και προϊόντα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για τις συγκεκριμένες εφαρμογές και τα προϊόντα και τις χρήσεις τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ισχύει και σε άλλες αντίστοιχες οδηγίες και για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και καλύτερη δυνατότητα ερμηνείας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα χρειαζόμαστε συγκεκριμένους ορισμούς ε, για τον κλάδο στο κείμενο. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η βελτίωση του ορισμού του περιεχομένου των ανακοινώσεων των ε, ε κρατών μελών για την κατάσταση της προμήθειας, της προμήθειας αερίου για τις συσκευές αυτές το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιούνται συσκευές αερίου σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις διάφορες ε, περιπτώσεις και να συμπεριλάβουμε και πολύ συγκεκριμένε απαιτήσει για τις ανακοινώσεις. χρειάστηκε να προσθέσουμε και κάποιες διατάξεις που διευκρινίζουν τη σχέση μεταξύ των συσκευών αερίου και του σχετικού κανονισμού με συγκεκριμένη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση. όσον αφορά τις άλλες ε, διατάξεις και τα άρθρα και τις συγκεκριμένες απαιτήσει, ε, θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να υπερβούμε το παρόν νομικό κείμενο, απλώς και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις για συντακτικές αλλαγές για βελτίωση της διατύπωσης και κωδικοποίηση και κάποιων πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται ε, από υπεύθυνου κατασκευαστές. Για παράδειγμα, υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση κινδύνου και γενικές αρχές σχεδιασμού στο παράρτημα 1, ε, που αφορούν τα ε, προϊόντα αυτά. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά το εύρος αυτού του κανονισμού, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να εντοπιστούν τομείς τους οποίους θα μπορούσε να επεκταθεί η ισχύ αυτού του κανονισμού παραδείγματος χάρη η χρήση του αερίου σαν καύσιμο δεν μπορούσε να γίνει με την έννοια, ε, επέκτες στον τομέα αυτό, με την έννοια ότι το θέμα της ασφάλειας ήταν ε, κάτι που μας ε, περιόρισε, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της υψηλής θερμοκρασίας στις εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα αυτά, στις συσκευές αυτές που χρησιμοποιούν ε, νερό. Υπάρχει το θέμα λοιπόν της υψηλής θερμοκρασίας του νερού και το θέμα της πίεσης. Σήμερα υπάρχει ειδική οδηγία που ορίζει τις ε, θερμοκρασίες και την ε, υψηλή πίεση στις συσκευές. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα μεταξύ των δύο αυτών κειμένων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καλυφθούν όλοι οι κίνδυνοι που προέρχονται από το αέριο, επίσης το πολύ σημαντικό θέμα της απόδοσης της ενέργειας, της χρήσης της ενέργειας στα πλαίσια αυτού του κειμένου και δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες καθότι υπάρχει νομοθεσία και νομοθετικά κείμενα που τίθενται σε ισχύ και αφορούν αποκλειστικά το θέμα της ε, ε, ενεργειακής ε, αποδοτικότητας. Θα ήθελα εδώ να σας δείξω ότι σε αυτή την δημόσια έρευνα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, υπέβαλαν προτάσεις και τροπολογίες, τις οποίες βεβαίως δεν θα σας τις ε, παρουσιάσω με λεπτομέρειες. Βλέπετε όλα τα σημεία εδώ, στα οποία καταλήξαμε. Περίπου τα 2 τρίτα ή τα 3 τέταρτα, δηλαδή περίπου 75-76% των απαντήσεων σε αυτή τη δημόσια μελέτη, είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών, τροποποιήσεων που προτείνουμε εδώ. Το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας, από τη στιγμή που εντοπίστηκαν οι ανάγκες, είναι να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα θέματα, συγκρίνοντας εναλλακτικές λύσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών στο νέο νομοθετικό κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς ότι το νομοθετικό πλαίσιο αυτό καθεαυτό θα παραμείνει αναλύωτο. Δηλαδή, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οι κατασκευαστές, οι ρυθμιστές, θα παραμείνουν οι ίδιοι στη διαδικασία. Στην πράξη λοιπόν εδώ πρόκειται για μία προσπάθεια αποσαφήνισης του νομικού αυτού κειμένου. Να είναι δηλαδή πιο ευανάγνωστο, πιο εύχριστο. Αλλά δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεν διευρύνουμε δηλαδή, αν θέλετε, τους τομείς εφαρμογής. Γι' αυτό και η μελέτη αυτή αξιολόγησης αντικτύπου καταλήγει στο ότι δεν υπάρχει σημαντική συνέπεια ακριβώς ε, εξαιτίας αυτού που σας ανέφερα. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλη αλλαγή στο νομοθετικό αυτό πλαίσιο. Εδώ βλέπετε τις διάφορες εναλλακτικές που εξετάσαμε και θεωρούμε ότι σαφώς θα πρέπει να συγκριθούν εδώ οι ποιοτικές πτυχές. Με την έννοια ότι δεν είδαμε ποσοτικές ε, αλλαγές. Για να τις συγκρίνουμε. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη είναι να μην κάνουμε τίποτα. Η δεύτερη είναι να παραμείνει το νομοθετικό κείμενο ως έχει και να βελτιώσουμε, να τροποποιήσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και η τρίτη ε, εναλλακτική είναι βεβαίως να αλλάξουμε το νομοθετικό αυτό κείμενο. 23 ερμηνευτικά κείμενα υπάρχουν ήδη, άρα βρισκόμαστε ε, ε, εκ των πραγμάτων ε, στην εναλλακτική λύση 2 και από ό,τι φαίνεται η σύγκριση των ποιοτικών επιπτώσεων είναι αυτών που πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στην αντιμετώπιση των αναγκών. Αποσαφήνιση λοιπόν του νομοθετικού πλαισίου. Αυτό επιλέγουμε. Θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στους στόχους μας, ενισχύει την ασφάλεια, ενισχύει την ε, ασφάλεια δικαίου, την εποπτεία, μια συνοπτική και συνεκτική προσέγγιση για όλους τους τομείς και φυσικά διευκολύνει και την εφαρμογή, την υλοποίηση. Τέλος, όπως και στις άλλες προτάσεις που έχουν υποβληθεί, διαπιστώνουμε ότι ο κανονισμός είναι το καλύτερο μέσο, το καλύτερο εργαλείο που ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εδώ. Κανονισμός, διότι με αυτό τον τρόπο πλησιάζουμε την απλοποίηση, δηλαδή έχουμε ένα νομικό κείμενο και όχι 29 μεταφορές ε, στην ομοθεσία των κρατών μέλων. Έχουμε λοιπόν μια πιο συνεκτική προσέγγιση και η νομική ασφάλεια ενισχύεται. Δεν μπορεί να υπάρξουν δηλαδή υπεραιτέρω διεκδικήσεις από μέρους των κρατών μελών και την ίδια ώρα όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας προσέγγισης παραμένουν. Οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προδιαγραφών προτήτων από τη στιγμή που συμμορφώνονται με τον κανονισμό θα παραμείνουν οι διαρθρώσεις ανατομέα, οι δυνατότητες συνεργασίας και θεωρούμε ότι εδώ δεν υπάρχει καμία απολύτως ε, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με την αρχή της επικουρικότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι διευκολύνουμε πολύ συγκεκριμένα και την υλοποίηση, την εφαρμογή και τις ε, εφαρμοστικές ε, διαδικασίες. Αυτή ήταν μια πολύ σύντομη παρουσίαση της αξιολόγησης αντικτύπου και κυρία Πρόεδρε ολοκλήρωσα την ε, παρουσίασή μου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Στάιλερ. Είναι η συγγήτρια, έχετε σχόλια, έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έτσι μπορώ και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά προηγουμένως να πω ότι το θέμα της προθεσμίας για μετάφραση, της ημερομηνίας για μετάφραση 20 Ιανουαρίου. Και θεωρώ πραγματικά ότι θα συζητηθεί στις 24 Φεβρουαρίου, άρα υπάρχει κάποιος χρόνος. Εμείς θέλουμε να έρθουμε σε επαφή βεβαίως ε, με τον κλάδο, με τους κατασκευαστές και οι σκιώδες και εγώ θα θέλαμε να διευκρινίσουμε κάποια σημεία με κάποιες ερωτήσεις. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, το θέμα της ε, παροχής αερίου, ιδιαίτερα διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν σήμερα νέες πηγές παραγωγής ε, αερίου. Το θέμα της απόδοσης λοιπόν των συσκευών είναι κάτι που δεν το είδα πουθενά και ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα. Μιλήσατε για την παροχή, για την προμήθεια αερίου, μιλήσατε για την εποπτεία της αγοράς, μιλήσατε για την εφαρμογή, για την υλοποίηση. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πραγματικά στην πρόταση αυτή μας απασχολεί η ασφάλεια των συσκευών αερίου, αλλά φυσικά μας ε, απασχολεί ιδιαίτερα και το θέμα της απόδοσης της ενέργειας όταν αγοράζουμε μια τέτοια συσκευή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 24 Φεβρουαρίου λοιπόν θα παρουσιάσω με πολλές λεπτομέρειες την έκθεσή μου, αλλά θεωρώ ότι πολύ σωστά θέσατε τα θέματα. Υπάρχει όμως ε, μεγάλη ευαισθησία και ανησυχία για το θέμα της ασφάλειας αυτών των συσκευών αερίου, γι' αυτό και επειδή και εμείς ε, εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε τη δική μας ε, ομάδα που ασχολείται με την αξιολόγηση αντικτύπου, θα είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με τα άλλα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, να δούμε ότι υπάρχει συνοχή μεταξύ όλων αυτών των προτάσεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας παρουσιάσετε και φυσικά θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας στα σημεία αυτά. Από το ΕΛΚΟ, κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ρουμανικά δεδομένου ότι πρόκειται για οδηγία τεχνικού ε, και βεβαίως θα περιμένω και την έκθεση της κυρίας Στήλε. Η οδηγία που αφορά τις ε, συσκευές αερίου είναι πάρα πολύ σημαντική και θέτει κανόνες αυστηρούς για την αγορά. Α, τις μελέτες είδαμε ότι ούτως ή άλλως μέχρι τώρα εφαρμόζεται σωστά αυτή η οδηγία, αλλά δεν μας λέει πώς θα πρέπει κάποιες ε, ε, κριτήρια και απαιτήσει να πληρώνται. Θα πρέπει πάντα να δίδονται οι σωστές τεχνικές λύσεις ώστε να διευκολύνεται η κατάσταση και να υπάρχουν κριτήρια εναρμονισμένα στην αγορά για θέματα ασφαλείας. Πράγμα το οποίο γινόταν μέχρι τώρα σε θελούσια βάση. Από την ε, εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που με προσοχή, έχω να κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να μου πει μέσω συγκρίσεων των ε, συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε η Επιτροπή, η ευελιξία έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των καταναλωτών. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ασφάλεια και τι ε, προβλέπει να απαιτήσει ως κριτήρια πιο αυστηρά στο πρώτο ε, παράρτημα για να υπάρχουν οι συνθήκες ασφαλείας για όλους. Η Κομίσιο S&D. Δεν έχω κανέναν παρά μόνο τον ε, Πασκάλ εδώ. Ο Πασκάλ, τι έχει να πει εκ μέρους των Όχι. Όχι. Κάποιος άλλος πρώτα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ε, παρουσίασή της. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προσθέσω πολλά πράγματα. Το μόνο που περιμένω είναι να δω την έκθεση. Δύο σύντομα σχόλια, όπως προηγουμένως και με τις εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι για την εποπτεία της αγοράς καλό θα ήταν να περιλάβουμε ένα κεφάλαιο και Συμφωνώ ότι ο κανονισμός είναι καλύτερος από την οδηγία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε τον κανονισμό αυτό πολύ σύντομα να τον εγκρίνουμε και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία μεταξύ μας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Πασκάλ θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ Βίκη. Απλώς θέλω να πω ότι είναι η μέρα μου σήμερα. Τέλος πάντων, ε, περιμένω την έκθεση και εμπιστεύομαι απόλυτα την εισηγήτρια στην οποία αναθέσαμε την έκθεση αυτή για το θέμα αυτό το τόσο σημαντικό. Thank you. Άλισον, θες να πεις κάτι για το θέμα αυτό, για την αξιολόγηση επιπτώσεων, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα νέα μέλη της Επιτροπής ε, θα ακούσουν τι κάνει το τμήμα το δικό σας εδώ στο Κοινοβούλιο. Thank you very much. Ευχαριστώ για να εξηγήσω τι κάνει το τμήμα μας με τις αξιολογήσεις επιπτώσεων. Εμείς είμαστε το τμήμα εκ των προτέρων αξιολογήσεων επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συστηματικά ετοιμάζουμε μια αρχική εκτίμηση για τα μέλη, για τις αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με μια σύνοψη που δίνει λίγο το ιστορικό της πρότασης, όπως παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διευκολύνονται λίγο ε, τα μέλη για την εξέταση του θέματος. Δεν κάνουμε εκτίμηση της πρότασης. Εμείς εξετάζουμε την ποιότητα της αξιολόγησης επιπτώσεων, εξετάζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κατάλογο φυσικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Ε, Τώρα, κατόπιν τούτου, για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση επιπτώσεων μπορούμε να είμαι πολύ σύντομοι, διότι όπως εξήγησε σαφέστατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πιθανές συνέπειε είναι πολύ περιορισμένες λόγω τη περιορισμένης φύσης των αλλαγών που προτείνονται. Επομένως, η αξιολόγησή μα είναι ότι η αξιολόγηση είναι αντίστοιχη αυτού που προτείνεται. Κάποιες από τις βασικές ε, ε πτυχές οι οποίες είναι θετικές νομίζω είναι ότι ε, φάνηκε ότι ήταν αρκετά εκτεταμένη η ε, ε, εφαρμογή στα κράτη-μέλη και αυτό σε σχέση με άλλες εκτιμήσεις επιπτώσεων είναι πολύ θετικό και επίσης υπάρχει μια αναλυτική περιγραφή στη διαβούλευση στα κράτη-μέλη οπότε είναι εύκολο να καταλάβει κανείς από πού προέκυψαν οι διάφορες απόψει και επίσης τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής από σε κανονισμό παρουσιάζονται με πολύ ε, λογικό τρόπο. Οι αδυναμίες ε, που εντοπίζουμε δεν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ε, θα αναφερθώ εντάχει σε κάποιες από αυτές. Αφορούν κυρίως την ποιότητα της διατύπωσης. Υπάρχουν πολλές επαναλήψεις που ορισμένες φορές δυσχεραίνουν την κατανόηση χωρίς να μπορεί να διαβάσει κάποιος όλο το κείμενο. Ε, και τα προβλήματα, επειδή δεν είναι ακριβώς προβλήματα, πρόκειται απλώς για κάποια μικρό ε, θέματα που δημιούργησαν μια σύγχυση, υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ της βασικής έκθεσης και της ε, ε σύνοψης και αυτά νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με την ουσία της συγκεκριμένη εκτίμησης επιπτώσεων. Η διάκριση μεταξύ των δύο βασικών στοιχείων είναι ε, δύσκολη. Εμεί θεωρούμε ότι αυτή είναι η βασική κατάσταση. Οι διάφορε επιλογέ που έχουμε στη διάθεσή μα είναι περιορισμένε, αλλά δεν μπορεί κάποιο να διακρίνει και κάποια άλλη επιλογή μεταξύ του να μην υπάρξει καθόλου νομοθεσία και να υπάρχει νομοθεσία. Ε, ε, τα μόνα θέματα τα οποία θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαν ίσω να εξεταστούν λίγο περισσότερο είναι θέματα τα οποία αναφέρθηκαν στην εκ αξιολόγηση που είναι πάντα κάτι θετικό ε, της επιπτώσεων. Παίρνει στοιχεία από την ε, εκ αξιολόγηση. Εδώ υπήρχε εκ αξιολόγηση που δεν γίνεται πάντα και εκεί φάνηκε ότι το κόστος συμμόρφωση ήταν υψηλότερο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, για παράδειγμα αλλά αυτό προφανώς ε, ε, είναι με γνώμονα την αρχική οδηγία όταν τέθηκε σε εφαρμογή προκλήθηκε το περαιτέρω κόστος και αυτό που προτείνεται τώρα δεν ε, ε, ε, προϋποθέτει επιπλέον κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέραν του αρχικού. Γι' αυτό ακριβώς και η επίπτωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρείται ουδέτερη. Αν δείτε όμως την αρχική οδηγία, όταν εισήχθη δημιούργησε κάποια προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν νομίζω όμως ότι αυτό αφορά το παρόν πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώνοντας λοιπόν για αυτό το σημείο θέμα, ε, να πω ότι το ανέφερε και η συγγήτρια, Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι και για το απογευματινό θέμα, γιατί δεν θα είστε εδώ, δεν είναι εδώ βέβαια οι σκιώδεις ηγητές, ίσως θα πρέπει να, να επανέλθουμε. Να σταθείτε δύο λεπτά στην έκθεση του κυρίου Κάλλας και να μας παρουσιάσετε και την άποψή σας για την εκτίμηση επιπτώσεων εκεί. Λοιπόν, για το PPE νομίζω το πιο εύκολο για να το συζητήσουμε και για να βοηθήσω και στη συζήτηση είναι σε σύγκριση με αυτή την εκτίμηση επιπτώσεων για τις συσκευέ αερίου. Γιατί νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι η οδηγία PPE για τον ε, προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό διευρύνει το πεδίο εφαρμογή και περιλαμβάνει και άλλα προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται. Ενώ σε αυτή την περίπτωση στι συσκευέ αερίου δεν υπάρχει ε, κάποιο νέο προϊόν το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα συμπεριληφθεί εδώ. Ε, λόγω του ορίου των 105 βαθμών Κελσίου. Υπάρχουν κάποια προϊόντα λοιπόν εδώ, όπως για παράδειγμα γάντια, ε, τα οποία ε, καλύπτονται στην οδηγία για τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας που δεν καλύπτονταν με την παρούσα λόγω του πεδίου Δεν υπάρχει εδώ κατανομή ανάλογα με τους διάφορους ενδιαφορομένους, ενώ στη συγκεκριμένη εκτίμηση επιπτώσεων έχουμε στοιχεία και είδαμε αμέσως ότι συμμετείχαν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεισέφεραν στις προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την άλλη πρόταση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, ίσως θα μπορούσε να μα το διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έγινε. Ε, διότι θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε. Η άλλη διαφορά είναι ότι δεν υπήρχε επίσημη εκ των υστέρων αξιολόγηση τη οδηγία για τον προσωπικό εξοπλισμό. Ε, είχε μια, υπήρχε μια άτυπη εκ των υστέρων αξιολόγηση, ε, στην οποία βασίζεται εν μέρη εκτίμηση επιστώσεων, αλλά δεν υπήρχε εκ των υστέρων αξιολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτού βέβαια, αλλά ίσως θα έπρεπε να το αναφέρουμε για το μέλλον οι εκκρεμότητες τώρα για την αξιολόγηση επιπτώσεων για τον προσωπικό εξοπλισμό ε, η οποία ε, να πω ότι είναι μια καλή εκτίμηση επιπτώσεων απλώς σας αναφέρω κάποιες αδυναμίες που εντοπίσαμε που δεν υπήρχαν στην εκτίμηση επιπτώσεων για τις συσκευέ αερίου και ίσως θα μπορέσει να δώσει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε περαιτέρω σήμερα το απόγευμα. Το τελευταίο θέμα στην ε, πρωινή μερίσια διάταξη είναι η έκθεση του Ότμαν Κάρας ε, ε, για το, η καταλληλότητα και την αποτελεσματικά της νομιοθεσίας Refit. Θα του δώσω απευθεία το λόγο. Ε, είναι κάποιος άλλος εδώ. Όχι, ο κύριος Κάρας λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, αύριο η Επιτροπή θα υποβάλει και θα δημοσιεύσει την, θα γνωστοποιήσει την ε, έκθεσή της. Εμείς ε, εδώ απλώς καλούμαστε να υποβάλουμε μια γνωμοδότηση. Εγώ στην πρότασή μου για την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας Αναφέρομαι στις ε, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, τις εκτιμήσεις ε, από τις διαβουλεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είναι η εφαρμογή και η θέση σε ισχύ της νομοθεσίας ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά και έχω λάβει υπόψη μου όλο το πρόγραμμα καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. Πρόκειται για μία εξελίξει νομική διαδικασία, νομοθετική διαδικασία, η οποία φυσικά έχει ξεκινήσει σε πολύ ευρύτερο επίπεδο και για όλα αυτά τα θέματα από το 2004 μέχρι και ολοκλήρωση της ε, έρευνας έχουμε λάβει υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία. Εγώ σας προτείνω εδώ 11 συγκεκριμένα σημεία, επιμέρους σημεία, ε, παραδείγματο χάρη ε, θέμενη αξία στην οδηγία, στον κανονισμό. Θα πρέπει να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός και αυτό για κάθε προσπάθεια νομοθετικού κειμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμμόρφωση, η συμμόρφωση, το κόστος, που θα πρέπει να υπολογίζεται, καθώς και το κόστος του να μην κάνουμε τίποτα, το κόστος της μη δράσης. Ε, θα πρέπει επίσης να επαναργοποιήσουμε το εργαλείο αυτό που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να κινητοποιήσουμε διάφορες ρυθμίσεις ε, που αφορούν την ε, υλοποίηση, τη θέση σε ισχύ, το gold plating αν θέλετε, το, η επικάλυψη θα πρέπει να αποφευχθεί εδώ με την έννοια ότι για κάθε συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου και μια μελέτη κόστους ωφέλειας. Επίσης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των κατεξουσιαδότηση πράξεων, των επιπτώσεών τους και πιστεύω ότι και στο Κοινοβούλιο αλλά και στις πολιτικές ομάδες και στην Επιτροπή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζονται αρμόδιοι για την παρακολούθηση αυτών των πράξεων των κατεντολή πράξεων. Και θα πρέπει επίσης να υπάρχει επικοινωνία, διεύλος επικοινωνίας με την ε, Επιτροπή, διότι πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι κάποιες πολιτικές συμφωνίες μπορεί να χαθούν, να εξανεμιστούν στα πλαίσια αυτών των ε, κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Εθνική Συμφωνία για το 2004 για την καλύτερη νομοθετική διαδικασία θα πρέπει εδώ να ισχύσει έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών πληροφοριών όσον αφορά την θέση σε ισχύ των πράξεων αυτών. Εγώ προσωπικά και το έχω ξαναπεί είμαι υπέρ του να αναφέρουμε πάντα την εντολή και εδώ αναφέρομαι Timmermans kann diese unabhängige Beratungsgruppe nicht ersetzen. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαβουλεύσεις και να γίνεται εγκαίρος με διαφάνεια η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα πρέπει επίσης να έχουμε μία σίγουρη ε, μέθοδο παρουσίασης των απόψεων έτσι ώστε να προσέχουμε πάντα να ακούγονται και οι απόψεις της ε, μειοψηφίας 8 σημείο, το θέμα του κόστους και της εξοικονόμησης και του περιορισμού των δαπανών καθότι τα κράτη-μέλη εδώ καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το θέμα αυτό. 9. Το θέμα της βελτίωσης της ποιότητας των ακροάσεων. Αυτό είναι κάτι που το έχω πει. Χρειαζόμαστε πάντα μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. 10. Η Europe σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε εδώ κάτι το οποίο δεν είναι επίκαιρο. Αναφέρθηκα και προηγουμένως στον κατακαιρματισμό. Ο κατακαιρματισμός συνεχίζεται και θα πρέπει σαφώς να εγγυηθούμε εδώ με κάθε τρόπο τις ε, πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ε, ενιαία διάδοσή τους. Εντέκατο σημείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει εδώ ότι θα κάνει αξιολογήσεις και θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά η παρούσα, η σημερινή νομοθεσία εφαρμόζεται με ορθό τρόπο, όπως παραδείγματο χάρη η οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές. Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να πλήξει και να αποτελέσει στρέβλωση της ενιαίας αγοράς. Αυτές είναι οι προτάσεις μου και φυσικά όταν προετοιμάσω την ε, γνωμοδότησή μου θα συμπεριλάβω όλα αυτά τα σημεία. Ποιο είναι σκιώδη. Εγώ θα μιλήσω σουηδικά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Νότμαρ Καράς για τη γνωμοδότησή του. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει δέσμευση ότι θα προχωρήσει σε απλούστευση όλων των κανόνων που ισχύουν. Εγώ σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μου το έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα αυτό υπάρχουν ε, κάποιοι κανόνες, κάποιες ε, προδιαγραφές που δεν είναι πλέον ε, ρεαλιστικές σήμερα. Θα πρέπει να τις αλλάξουμε και για τις επιχειρήσεις και για τη χώρα γενικότερα. Και το κοινοβούλιο μας νομίζω ότι πρέπει να στείλει πολύ σαφές μήνυμα στην Επιτροπή. Είναι σημαντικό να ενεργήσουμε σωστά, διότι δεν θα πρέπει οι παρερμηνίες να δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα λειτουργίας. Εγώ ξέρω πως έχει η οργάνωση σε τέτοιου θέματα στην Σουηδία και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκητης και πορές φορές ξέρουμε ότι τα λόμπι ασκούν πιέσεις και η νομοθεσία και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται πολύπλοκη και αναποτελεσματική. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσωπικοί. Κατά την άποψή μου το REFIT είναι πάρα πολύ χρήσιμο διότι θα απλουστευτούν κάποιες διαδικασίες, αλλά να μην το πολιτικοποιήσουμε το όλο θέμα. Θα πρέπει να ενεργήσουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχουμε καλύτερη ποιότητα και πιο αποτελεσματική και να προβλέπουμε κανόνες και προδιαγραφές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και ρεαλιστικά. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την αγορά και τους εργαζόμενους αν θέλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και πιο παραγωγικοί με κατάλληλη νομοθεσία. Η θωράκιση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και δεν θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε έχοντας υπόψη μόνον τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, διότι έτσι θα κάνουμε στο τέλος κάτι το οποίο θα είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Η συνεργασία μας όντως νομίζω ότι θα είναι καλή, αλλά Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να προσέξουμε δεδομένου ότι στο κείμενο υπάρχουν πάρα πολλά κενά και δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε να περάσουν. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, κάποιοι κανόνες τους οποίους μπορούμε να πλουστεύσουμε, να διαγράψουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε και αναπροσαρμογή κάποιων κειμένων, διότι είναι δικό μας θέμα τελικά η προστασία του κατανοτού και θα πρέπει να την κάνουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Could somebody please, taking a list of speakers? Θέλετε παρακαλώ από τη γραμματεία να ε, σημειώσετε ονόματα των συναδέλφων που θέλουν να λάβουν το λόγο. Εκ μέρους της ECR, εγώ είμαι η σχέση συγγετρία, θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ασχολείται με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και στο σχέδιο γνωμοδότησή σας, πολλά τα οποία είπατε με βρίσκουν σύμφωνοι, κυρίως όσον αφορά τη μιμία, πρώτα απ' όλα την απλούστευση, το θέμα της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, τα θέματα καταβολής κάποιων επανών, Πολλά κοινά στοιχεία έχουμε. Τώρα, πρέπει να πω ότι εχθές, ε, Επιτροπή το θέμα του Refit συζητήθηκε και είπαμε ότι χρειαζόμαστε όχι μόνο νέα νομοθεσία, αλλά να δούμε και αν ήδη η κείμενη νομοθεσία είναι η καταλληλότερη και πιο αποτελεσματική. Διότι από την αρχή ε, της προπαρασκευαστικής εργασίας μέχρι την ε, εφαρμογή της και την ε, παρακολούθηση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η ομάδα μου πιστεύει ότι θα πρέπει να δούμε όλοι λοιπόν την εργασία, την διαδικασία αν θέλετε από το στάδιο της προπαρασκευαστικής μέχρι της εφαρμογής επαναλαμβάνω. Είχαμε κάποιες ε, ιδέες όσον αφορά τις ε, διάφορες ε, ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, δηλαδή πρέπει να εξισορροπήσει κάπως η νομοθεσία αν θέλετε. Βάζετε κάτι το οποίο είναι πιο σύγχρονο, αφαιρείτε κάτι το οποίο είναι παλαιωμένο. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να προσπαθήσουμε να κάνουμε και κυρίως να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει την Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική. Θα πρέπει πάντα, ό,τι και να κάνουμε, να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και σε ποιους τομείς και εκτός Ευρώπης. Θα πρέπει επίσης να είναι όσοι ασχολούνται με την εκτίμηση επιπτώσεων να το κάνουν αυτό μέσα σε ένα πνεύμα ουδετερότητος, διότι δηλαδή πολλές φορές στο παρελθόν ότι Φτάνει η εκτίμηση επιπτώσεων στην Επιτροπή και πολλές φορές ε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να πει ούτε η εκτίμηση ούτε η Επιτροπή εκ των υστέρων. Καλό θα ήταν να είχαμε και εμείς την μονάδα μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει τέτοιου είδους εκτιμήσεις με ανεξάρτητο τρόπο. Τώρα, εξαιρέσεις, θέματα που αφορούν τις ΜΜΕ είναι σημαντικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης για το θέμα αυτό, για τις ΜΜΕ, το σύνολό τους, ώστε να μπορούμε να ενεργήσουμε στους τομείς που πιστεύουν εκείνοι ότι είναι προτεραιότητας με διαβουλεύσεις Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε και καλύτερη νομοθεσία ε, σε θέματα κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις και θα πρέπει να τις εξετάζουμε εκ των προτέρων πολύ καλά πριν να προχωρήσουμε στην επιλογή και εφαρμογή τους. Θα πρέπει πάντα να κάνουμε την σωστή αξιολόγηση και να μειώσουμε το άχθος. Πολλά έγιναν στην προηγούμενη φοιτεία για το θέμα αυτό του κανονιστικού πλαισίου και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι έχει γίνει στο θέμα αυτό μέχρι τώρα και να ξαναρχίσουμε από την γραμμή από την Αθή. Υπάρχουν ήδη κάποια θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει και με τον εισηγητή σε θέματα με νομοθεσία η οποία έχει περάσει. Τι γίνεται εκ των υστέρων. Θα πρέπει να ξέρουμε αν πραγματικά από την ε, θεωρία έχει περάσει σωστά στην πράξη εφαρμογή της και μαζί με τους άλλους συναδέλφους και εγώ θα ήθελα να θέσουμε κάποιες τροπολογίες πριν να εκπνεύσει η προθεσμία. Κυρία Ολατόμα, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική, συνοπτική και συγκεκριμένη γνωμοδότησή του, όντως θα πρέπει να δούμε από την νομοθεσία τι σημαίνει για τις μιμιέ η απορρίθμιση της νομοθεσίας, διότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι ο κεντρικός ιστός της Ευρώπης και της αγοράς εργασίας γενικότερα. Και όλοι προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά να έρθουν οι επιχειρήσει πίσω στην Ευρώπη, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και εγώ είμαι πεπισμένη ότι η απορρίθμιση για τις ΜΜΕ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης που είναι τόσο σημαντικέ για αυτές. Επίσης πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, οι ενεχόμενοι σε τέτοιου είδους θέματα και στην μελλοντική μας εργασία θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η δική τους άποψη επί του θέματος αυτού. Επίσης, συμφωνώ με αυτά τα οποία τονίσατε, ότι είναι απαραίτητο να μην έχουμε υπερβολική νομοθεσία και κανονισμούς, να μην υπερθεματίζουμε σε τέτοιου θέματα. Υπάρχουν εδώ κάποιοι εκπρόσωποι ΜΜΕ εδώ, οι οποίοι ακούνε τι λέμε. Και προηγουμένως τους ρώτησα ποιες είναι οι δικές σας ε, ε, προτεραιότητες κατά την απόψη μας. Είπαν τρεις είναι. Πρώτα απ' όλα. Deregulation, deregulation, deregulation. Κατάλληλη νομοθεσία, πλούστευση της νομοθεσίας. Και ο κύριος Τίμερμανς που ασχολείται με το άλλο θέμα. Ελπίζω ότι θα μας εκπλήξει θετικά, διότι αυτό είναι το θέμα του. Θα πείσω ότι το θέμα του, του της καλύτερης νομοθεσίας και της απλούστευσης της ε, των λιγότερων κανονισμών να μας βοηθήσω και προστρέχω σε πολύ θετική συνεργασία με τον εισηγητή το οποίο περιμένουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο Ντένις Τιγιάνγκ δεν είναι εδώ. Ε, κύριε Μαστάλκα, αντικαθιστάτε τον Ντένις, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης ηγητής βέβαια, αλλά συμμετέχω στην Επιτροπή. Επομένως, ε, με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό που παρουσίασε εδώ ο κύριος Κάρας. Στην ε, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα προσπαθήσω να τα παρουσιάσω αυτά, διότι για μας αυτό αποτελεί θέμα προτεραιότητας. Όταν ακούσαμε την Επίτροπο Γιούροβα, ε, τη ρώτησα ειδικά ε, μια ερώτηση για το Refit, διότι θεωρώ ότι αποτελεί προτεραιότητα και θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία ε, για το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για τον ε, πολύ συγκεκριμένο τρόπο ε, με τον οποίο μας παρουσίασε τα πράγματα ο κύριος Κάρας. Έχει μιλήσει με ενώσεις επιχειρήσεων ε, και με τον πρόεδρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να πω το εξή. Όλα αυτά δεν θα μας οδηγήσουν πουθενά αν έχουμε μελέτες σαν αυτή που είδαμε απλώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προηγουμένως, όπου ε, το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, που ρωτήθηκαν ήταν κάτω από το 40%. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια αποτελέσματα ε, σε μελέτες επιπτώσεων. Έχουμε 99% μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, έχουμε μελέτες τις οποίες δεν αναπαντούν. Αυτές οι μελέτες είναι άχρηστες στην πραγματικότητα. Ε, αν θέλουμε πραγματικά να μελετήσουμε πώς λειτουργεί ο κλάδος, θα πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά ανάλογα και με τη συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, ένα ποσοστό το οποίο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Small Business Act είναι στην πραγματικότητα θεωρία σε πολλές χώρες το γενικό γεγονός ότι δεν γίνεται καμία δοκιμή για να ε, δούμε πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία. Συμμετείχα και εγώ σε κυβέρνηση και ξέρω ότι ε, υπήρχαν συνεχώς ε, φόροι επιφόρων και στο τελευταίο διάστημα στο οποίο ήμουν υπουργός κατάφερε να περάσει ένα νόμο ο οποίος έλεγε ότι οποιοδήποτε επιπλέον κόστος, οποιαδήποτε επιπλέον φορολόγηση θα πρέπει να περνάει και από το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να μπορεί να γίνει μια μελέτη των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε νέα φορολογία. Αντί λοιπόν να πηγαίνουμε προς περαιτέρω απορρίθμιση, ε, ε, προσθέτουμε επιπλέον νομοθεσία και επιπλέον κανόνες. Και όπως έλεγε και ο ε, εισηγητής, υπάρχει πάρα πολύ νομοθεσία και κανονισμοί. Είναι όλα υπερβολικά αυτά. Αν μπορέσουμε λοιπόν να εξετάσουμε κάθε φορά το κόστος της νομοθεσίας ή της μη εφαρμογής νομοθεσίας, τότε θα μπορούμε να διαμορφώνουμε συγκεκριμένη άποψη. Αλλιώς οι ε, μικρόσες επιχειρήσεις δεν θα βοηθούνται από αυτό που κάνουμε, απλώς ε, θα τους χρυσώνουμε το χάπι. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν και ελπίζω εμείς από την Επιτροπή μας να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, σε κάτι απτό το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει το πρόβλημα να αντιμετωπίσει και εγώ ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μου απάντησε τίποτα. Εγώ που ε, τι ρώτησα. Ε, η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγμή. Τι νέα μέτρα θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά για την νομοθεσία αυτή, την οποία θέλουμε να τη βελτιώσουμε ή τη θέλουμε να την θέσουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις and welcome to the SMEs at the back of the room. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κάρας για την εξαιρετική του και πολύ σημαντική εργασία. Φυσικά και το θέμα αυτό αφορά μέσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται τα αποτελέσματα, θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά την ορολογία που χρησιμοποιείτε, Απορρίθμιση λέτε. Όχι, δεν πρόκειται για απορρίθμιση. Πρόκειται για μια καλύτερη νομοθεσία και ρύθμιση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί η απορρίθμιση ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει σε 28 διαφορετικές ρυθμίσεις Δηλαδή στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από το, το οποίο θέλουμε να φτάσουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να το προσέξουμε και να βρίσκεται στην καρδιά των ε, προσπαθειών μας. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι από την πολιτική μας ομάδα. Το θέμα τώρα της αξιολόγησης. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε η αξιολόγηση αντικτύπου θα πρέπει να γίνεται, είναι κάτι πολύ θετικό, αλλά θα πρέπει να γίνεται με ουδέτερο τρόπο, με αντικειμενικό τρόπο, γιατί οι κανόνες και οι ρυθμίσεις που προετοιμάζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν μόνο σκοπό να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις, αλλά και τους πολίτες. Η αξιολόγηση λοιπόν αντικτύπου θα πρέπει να στοχεύει και την ε, έρευνα στον τομέα της καθημερινής ζωής των πολιτών μας. Τι αλλάζει, τι επιπτώσεις υπάρχουν, ναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι για την οικονομία, αλλά σας παρακαλώ ας προσέξουμε λίγο και την κοινωνία, τους πολίτες, τους καταναλωτές. Και νομίζω ότι εδώ κάτι παραπάνω θα πρέπει να κάνουμε. Ένα τρίτο σημείο. Κύριε Κάρας. Εδώ έχω πρόβλημα με το κείμενό σας. Έχω την εντύπωση ότι δεν το θέλετε, αλλά χωρίς να το θέλετε, δίνετε την εντύπωση, τουλάχιστον εγώ αποκόμισα αυτή την εντύπωση, ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να θεσμοθετηθεί λίγο η διαδικασία για την εμπλοκή των ε, ενδιαφερόμενων φορέων. Εγώ εδώ λίγο δυσκολεύομαι. Ξέρετε ότι οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι ε, φορείς, οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν τελείως διαφορετική, αν θέλετε, ισχύ και θέση ανάλογα με την οικονομική τους καταρχήν δύναμη. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ιδιαίτερα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ένας μεγάλος βιομηχανικός σύνδεσμος καταλαβαίνετε ότι πολύ πιο εύκολα μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες από κάποια πολύ μικρότερη ε, οργάνωση προστασίας του περιβάλλοντος ή προστασίας των καταναλωτών. Είναι θέμα ισχύως και προτείνω εδώ να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στο κείμενό σας. Σόλτες besedo. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι φυσικά εμείς οι πράσινοι δεν ε, είμαστε αντίθετοι με τις προτάσεις αυτές. Θα θέλαμε όμως να γίνουν κάποιες προσθήκες. Συμφωνούμε όσον αφορά την απλοποίηση. Απλοποίηση, απλοποίηση, απλοποίηση, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθότι πολλές φορές σε εθνικό επίπεδο ακούμε ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις και νομοθετικά κείμενα. Όμως η απορρίθμιση, deregulation, επίσης έχει αρνητικές συνέπειες απλοποίηση που οδηγεί στην απορρίθμιση είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε. Και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε την απορρίθμιση, προσέξτε μην περιορίσουμε κάποια σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα, όπως όσον αφορά από τα επιδόμετα ανεργίας, παραδείγματο χάρη, την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, τα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την ε, διατροφική ασφάλεια, στον τομέα των τροφίμων. Πιστεύω λοιπόν ότι στην γνωμοδότησή μας θα πρέπει να είμαστε πολύ ισορροπημένοι όσον αφορά την απαραίτητη ρύθμιση και νομοθεσία που χρειαζόμαστε και την απλοποίηση που είναι επίση απαραίτητη. Στο σημείο 6 έχω ένα συγκεκριμένο σχόλιο. Ο εισηγητή αναφέρθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς. Εδώ δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους καταναλωτές, τις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σαφώς και θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και ένα τελευταίο σχόλιο επιτρέψτε μου. Όταν γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου, όταν κάνουμε μια τέτοια αξιολόγηση επιπτώσεων, είναι πολύ σημαντικό το ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγονται. Τα ορθά κριτήρια είναι καθοριστικά έτσι ώστε αυτή η αξιολόγηση επιπτώσεων να φτάσει σε σωστά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν στοχευμένη νομοθεσία, ορθή νομοθεσία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταπατήσουμε θεμελιώδη δικαιώματα ή να παραβιάσουμε σημαντικά και εκτιμένα δικαιώματα. Η Κάθριν Στάιλερ. Μετά ο κύριος Κάρας και τελειώσαμε. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη αυτό. Ακούγοντας τους συναδέλφους, διαπιστώνουμε ότι η έννοια την οποία συζητούμε, το gold plating, δηλαδή η υπερβολική ρύθμιση, η υπερβολική κανονισμή είναι κάτι που σίγουρα μπορεί να οδηγήσει σε μία επιστροφή σε εθνικές ε, ε, αντιμετωπίσεις. Και βλέπουμε την ε, δυσφορία που γεννιέται σε κάποια κράτη-μέλη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζουν λοιπόν αυτές τις προτάσεις και είναι σημαντικό όταν προχωρήσει αυτό το κείμενο να υλοποιηθεί. Βέβαια δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί, να τεθεί σε ισχύ πριν ε, ψηφιστεί αλλά ας προετοιμάσουμε καλά το κείμενο, ας δούμε στην πράξη ποια είναι αυτά τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στο κείμενο αυτό και ας ε, αποφύγουμε την υπερβολική νομοθεσία γιατί βεβαίως το είπατε και εσείς υπάρχουν τόσο πολλά άλλα νομοθετικά κείμενα τα οποία υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποίο όμως βλέπουμε ότι όταν ε, πρέπει να εφαρμοστούν στα κράτη-μέλη, προσκρούν σε σημαντικές δυσκολίες. Φυσικά λοιπόν, για να αποφύγουμε τις 28 διαφορετικές νομοθεσίες, γιατί αυτό είναι και ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουμε στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να προσέξουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για την εργασία που κάνατε μέχρι τώρα και εγώ συμφωνώ ότι όταν μιλάμε για εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλες ομάδες συμφερόντων και ε, φορείς εκτός των επιχειρήσεων. Πρόεδρος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό πάντα να ξεκινάμε από το υπάρχον ε, νομοθετικό καθεστώς από το status quo και γι' αυτό και θεωρώ ότι επειδή ακριβώς όλοι μας περιμένουν και μας παρακολουθούν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να κινητοποιήσουμε τους πολίτες και να δημιουργήσουμε διάλογο είναι καλό. Ο κύριος Κάρας, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Ήταν όλα πολύ επικοδομητικά τα σχόλιά σας. Τίποτα δεν ε, ακούστηκε που να αντιτίθεται σε όλα αυτά που προτείνω και πραγματικά αυτά που ακούσαμε είναι παρατηρήσεις για περισσότερη διευκρίνηση και αποσαφήνιση. Το θέμα της απλοποίησης απορρίθμισης δεν θα πρέπει αυτές οι δύο έννοιες να είναι αντίθετες. Χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθετική ρύθμιση, καλύτερη διακυβέρνηση. Με ποιο τρόπο, με ποια εργαλεία και απορρίθμιση σε καμία περίπτωση δεν είναι επιστροφή στις εθνικές ε, νομοθεσίες. Έχουμε την κοινοτική, την ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία πρέπει να βελτιωθεί, η οποία πρέπει να είναι η βέλτιστη. Και γι' αυτό και αυτή η απλοποίηση θα πρέπει σαφώς να έχει σαν σκοπό σε καμία περίπτωση την, ε, σε κάθε περίπτωση επιστροφή στην εθνική νομοθεσία, αλλά την καλύτερη νομοθεσία. Φυσικά και δεν εννοούσα, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που ακούστηκε, ότι θα πρέπει να ακουστούν μόνο οι απόψεις των επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές, οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες φυσικά θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης. Τρίτο σημείο, τρίτο τομής, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι, αν θέλετε, πιο θεσμοθετημένη συμμετοχή τους. Σε καμία περίπτωση δεν είχα την πρόθεση να περιορίσω τη συμμετοχή. Ε, θεωρώ ότι η συμμετοχή όλων των κατηγοριών φορέων είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όλοι πρέπει και μπορούν να συνεισφέρουν για να είναι πλήρης αυτή η αξιολόγηση. Και τέταρτο σημείο είναι η διευκρίνηση, η αποσαφήνιση κάποιων σημείων. Θα περιμένω όλες σας τις προτάσεις, κάποιες έχουν ήδη υποβληθεί σαν τροπολογίες, αλλά σκοπός μας είναι βεβαίως να συνεχιστεί η διευκρίνηση και αποσαφήνωση όλων των ενιών και προσβλέπω σε μια θετική συνεργασία, επικοδομητική συνεργασία μαζί σας. 10 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή και όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εξαιρετική συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε το απόγευμα.